Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινήσουμε. Δύο θεματικά έγγραφα έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Ζητώ συγγνώμη που αργήσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά είχαμε διάφορα εκρεμή ζητήματα να λύσουμε. Έγγραφο εργασία λοιπόν υπαριθμών 6 το πρώτο Ευρωπαϊκή Οικονομία για Βιομηχανία αντιμετώπιση με την κλιματική αλλαγή συναρμόδιος θεματικός συντονιστής ο κύριος Άικχαουτ είναι εκείνος ο οποίος θα μας κάνει την παρουσίαση του εγγράφου για να το συστήσουμε. Παρακαλώ. Κύριε Άικχαουτ. Α, θα αλλάξω στη μητρική μου γλώσσα τα Ολλανδικά και θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για μένα. So you can all Οπότε ετοιμαστείτε, φορέστε τα ακουστικά σας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έγγραφο είναι σαφές ότι έχει σαν πρόθεση να διευρύνει το πεδίο των συζητήσεων για την κρίση. Διότι θα υπάρξουν και άλλες κρίσεις στο μέλλον. Η κλιματολογική κρίση επαναλαμβάνεται, αναφέρεται περισσότερο από μια φορά, αλλά έχουμε και την ε, κρίση στον τομέα των τροφίμων όπως είναι η έλλειψη ε, ύδατος επίσης και πρώτων υλών επίσης ε, η έλλειψη, όπως είναι τα μέταλλα. που περνούν και αυτά και πρώτες ύλες και τα μέταλλα κρίση. Δεν είναι σαν να έχουμε μόνο μία κρίση και αν τη λύσουμε ε, ξεπερδέψαμε. Θα υπάρξουν πολλές κρίσεις στις επόμενες δεκαετίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ό,τι και να γίνει θα χτυπήσει και τον αριθμό των 9 δισεκατομμυρίων ο παγκόσμιο πληθυσμό. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ανάπτυξη, θέλουν ε, μάρια, θέλουν ε, τροφή, θέλουν ε, ένδυση και θέλουν και τις ανέσεις που απολαμβάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον, προς ένα πληθυσμό 9 δισεκατομμυρίων και να λάβουμε υπόψη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν πόρους. Βλέποντας το μοντέλο της καταναλώσεως ε, βλέπετε ότι βάζουμε μεγάλο βάρος, τεράστιο βάρος στον ε, πλανήτη και δεν είναι μόνο θέμα ενέργειας. Πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την ενέργεια και λέμε ότι τα προβλήματα είναι μόνο στην ενέργεια. Αλλά ε, να χρησιμοποιούμε πιο την ενέργεια και να μην εκπέμπονται πολλά αέρια του άνθρακος. Αλλά νομίζω ότι το δίκτυο μας πρέπει να γίνει μεγαλύτερο, να, να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή διότι υπάρχει και πρόβλημα σπάνιδος ύδατος σε πολλά μέρη του κόσμου. Ε, και επίσης ε, και γεωργική παραγωγή σπανίζει και αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη βιοπικιλότητα ε, θα πρέπει θα περιοριστεί και ο χώρος και το έδαφος που καλλιεργείται για την παραγωγή προϊόντων για κατανάλωση. Εντάξει, δεν απλώς μια ομιλία πρασίνου, παρόλο που είμαι πράσινος, αλλά μιλούμε και για, για γεωπολιτικές εντάσεις που δημιουργηθούν από όλα αυτά. Αρχίζουμε και το βλέπουμε ήδη. Όσον αφορά την έλλειψη γεών, την έλλειψη νερού, αυτά τα προβλήματα θα επιδεινωθούν στο μέλλον, δεν θα βελτιωθούν. Υπάρχουν κάποια μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στους φορητούς υπολογιστές και στα έπιπλα 95% από αυτά που παράγονται, προέρχονται από την Κίνα, από αυτά που καταναλώνουμε. Και αν καταναλώνουμε παρόμοια παρεμφερή προϊόντα περισσότερα, όλο και περισσότερο θα εξαρτώμαστε από άλλες χώρες του κόσμου, άλλα μέρη του κόσμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να γίνει αυτάρκης σε κάποιες πρώτες ύλες και πώς θα χρησιμοποιήσει σωστά ε, τους φυσικούς της πόρους η περιβαλλοντικά φιλική οικονομία δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι κάτι σημαντικό και ουσιώδες. Πρέπει να γίνουν πολιτικές επιλογές βέβαια. Πρέπει να δούμε τα, τα διάφορα προγράμματα των διαφόρων ηγετών. Θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα, ναι ή όχι. Αυτές είναι οι επιλογές που πρέπει να γίνουν. Ε, αφού ξέρουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων. Νομίζω ότι έχουμε μια δυνατότητα στην Ευρώπη και να γίνουμε ανταγωνιστικοί παρά αυτούς τους περιορισμούς. μιλάμε για βιωσιμότητα όσον αφορά την ενέργεια και τη μετώπιση της αλλαγής του κλίματος. δεν απλώς θέση των πρασίνων. Πρέπει να αλλάξει η πορεία η οικονομία μας δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις συνήθες διαδικασίες με μια απόχρωση πράσινη απλώς. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Όπως βλέπετε στην έκθεσή μου, μιλώ και απο, για αποδοτική χρήση των πόρων. Δηλαδή μια οικονομία που χρειάζεται λιγότερη εισρωή πρώτων υλών. Δεν μπορούν όλα να είναι συνάρτηση του ΑΕΠ και αυξήσεως της παραγωγής και μεγαλύτερης κατανάλωσης. η οικονομία μας βασίζεται σε αύξηση όλων αυτών των παραγόντων. Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε πιο αποδοτικοί όσον αφορά τη χρήση των φυσικών μας πόρων. Η παραγωγή μας χρησιμοποιεί λιγότερους φυσικούς πόρους, να είναι πιο αποδοτική. Και αυτή είναι μια θεμελιώδης αλλαγή της προσέγγισης όσον αφορά την οικονομία. Αυτό αναφέρει η έκθεσή μου. Αναφέρομαι στο ότι λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την προσέγγιση του ΑΕΠ δηλαδή οικονομία βάση αναπτύξεως στο ΑΕΠ και μόνο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων. Ε, είμαι περίεργος να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις σας. Εγώ έχω υποβάλει πρακτικές προτάσεις και λέω ότι πρέπει να έχουμε μια αλλαγή της προσέγγισής μας. Να δούμε και πώς λειτουργεί και το σύστημα εμπορίας ρήπων. Σκοπός αρχικά ήταν να δοθούν κίνητρα για τη μείωση εκπομπών του διοξιδίου του αλλά με την πάνω του χρόνου η πρακτική εφαρμογή του μέτρου οδηγεί στο να μην πετυχαίνουμε αποτελέσματα όσον αφορά τις τιμές. Να μην πετυχαίνουμε τους στόχους που είχαμε. Οι στόχοι ίσως να μην υπήρχαν σαφείς. Έχουμε, οι τιμές δεν μειώθηκαν αρκετά όσο θέλαμε. Και δεν νομίζουμε ότι, ε, δεν νομίζω ότι μόνο οι δυνάμεις της αγοράς θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε την απαραίτητη καινοτομία που είναι τόσο σημαντική για το μέλλον. Θα πρέπει να καθοριστεί σωστή τιμή όσον αφορά το σύστημα εμπορίας ρήπων. Να δώσουμε πραγματικά κίνητα στην αγορά, να, να προσελκύσουμε μάλλον επενδύσεις ε, για πράσινη τεχνολογία, για αποδοτική χρήση της ενέργειας. Η ενεργητική αποδοτικότητα θα είναι βασικό στοιχείο να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια. Γι' αυτό παράγουμε και να ανοίγουμε, δημιουργούμε ευκαιρίες για καινούριε εταιρείε που να μπορούν να επενδύσουν σε ε, τεχνολογία που χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Αλλά πρέπει να θέσουμε και δεσμευτικού στόχους ούτω ώστε να ξέρουν όλοι ότι είμαστε σοβαροί όταν θέτουμε τους στόχους, ότι το εννοούμε. Ε, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να διστάσουμε θα πρέπει να είμαστε δραστήριοι. Αυτό λέω. Πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό έχει και επίδραση στο φορολογικό σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια φορολογική ανταμοιβή για τη σωστή συμπεριφορά, για την καλή συμπεριφορά. Για να υπάρχει μια πίεση για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους πίεση πρέπει να έχουμε. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία συνάμα για να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε με κάποια συνέπεια. Προχωρώντας, Πρόεδρε, εν κατακλείδη, θέλω να πω ότι σκόπιμα διεύρυνα την, ε, το πεδίο που καλύπτει η συζήτησή μας. Δεν μιλώ μόνο για την αλλαγή του κλίματος. Ήθελα να ρίξω το δίχτυ μου πιο απλωτά, να καλύψω περισσότερα θέματα για να χρησιμοποιούμε καλύτερο τρόπο τους φυσικούς μας πόρους. Αυτό έχει συνέπεια για τη γεωργία, για την πολιτική για το νερό, και θα είναι στο επίκεντρο της μελλοντική οικονομικής μας προσέγγισης. Και σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ε, με τις πολιτικές επιλογές που απαιτούνται. Εγώ προσπάθησα να αναφέρω ποιε είναι οι επιλογές. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι προοδευτική, ότι προηγούμεθα στο παιχνίδι, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, οι θα εφαρμόσουν οι εταίροι μας πιο αποδοτική οικονομία και εμείς θα κυνηγάμε να τους στάσουμε. Πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Ηγέτες και όχι ουραγοί. Αυτή είναι η εισαγωγή μου και σας ευχαριστώ Πρόεδρε και όλους τους άλλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να σχολιάσουν. Η έχεις το λόγο Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, συμβολή Νομίζω ότι τα θέματα αυτά δεν βρίσκονται μένουν στο επίκεντρο της κρίσης. Παρ' αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν τόσο στη διάγνωση, στο επίπεδο της διάγνωσης, όσο και στη χάραξη στρατηγικής που προτείνουμε για να εξέλθουμε από την ίδια την κρίση. Όταν ε, προσεγγίζουμε όλα αυτά τα θέματα, θα ήθελα να πω ότι δεν αντιστέκομαι στην ανάγκη, ε, στην διαπίστωση της ανάγκης να διαρωτηθούμε για τους ίδιους μας αυτού. αυτούς. Την εποχή πριν από την κρίση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ε, Γερμανική Προεδρία το Μάρτιο του 2007 όρισε αυτό που για μένα είναι η η καρδιά του περιεχομένου αυτής της ε, στρατηγικής και έκανε την σωστή διάγνωση εν σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης για το 2020. Η δυσκολία είναι να δούμε κατά πώς τα συμπεράσματα τα οποία αντλήθηκαν από αυτή τη διάγνωση και από αυτή την στρατηγική που ορίστηκε επακριβώς μεν και σωστά ήταν τα σωστά. Και νομίζω ότι εδώ η έκθεσή μας μπορεί να δώσει μια σημαντική συμβολή. Γιατί αυτό το οποίο έγινε μέχρι στιγμής ήταν ε, το λεγόμενο νομοθετικό πακέτο κλίμα και ενέργεια που είναι ένα πακέτο ορισμού του πλαισίου της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτό. Και αυτό το οποίο μας λείπει είναι οι επενδύσεις, οι άμεσες επενδύσεις σε μια χρονική συγκυρία που γνωρίζουμε ποιο είναι το δημόσιο χρέος των χωρών μελών και που οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι τόσο ενεργές. Εάν θέλουμε να ελοπίσουμε αυτή την ημερήσια διάταξη στο πρόγραμμα, έχουμε ανάγκη ενώ μια δημόσιας επένδυσης όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πλήρω το ρόλο της μέσω των ευρωομολόγων και μέσω μηχανισμών που ήδη είχαμε την ευκαιρία να αναφέρουμε. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποιες ιδέες όπου η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεσο τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερως χρήσιμη. Και αναφέρω ως παράδειγμα ε, την ε, εκπόνηση ενός, ε, τη σύσταση ενός δικτύου, μιας δικτύωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και ξέρουμε τι γίνεται με, όταν καλούνται οι εταιρείε να το κάνουν. Πολλές φορές χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια και χρειάζονται και ενδιάμεση. Ε, η Επιτροπή θα πρέπει να ε, θεωρεί ως, τον εαυτό της ως υπεύθυνο για τον ορισμό μιας τέτοιας στρατηγικής. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του, της τιμολόγησης, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε, γιατί θα πρέπει να δώσει κίνητρο για επένδυση η τιμή και θα πρέπει να είναι αποτρεπτική για τους καταναλωτές και θα πρέπει να είναι ε, σωστή για να μην δημιουργήσει ενεργειακή ένδια. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μόνα τους. Χρειάζεται μια ρύθμιση της τιμής της ενέργειας που θα πρέπει κάποια στιγμή να τη δούμε εκ του σύνεγγης. Και δεν θέλω να με ακρηγορήσω. θα ήθελα να φέρω δύο ακόμα ιδέες. Η πρώτη είναι να επαληθεύσουμε με τον θεματικό μας εισηγητή εδώ ε, πώς θα αντιδράσουμε μια ιδέα που συζητιέται ευρέως, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του εφοδιασμού με τρίτες ε, δυνάμεις. Ξέρετε ότι η Ένωση ως ενεργειακή κοινότητα θα πρέπει να διαπραγματευτεί τον εφοδιασμό σε αέριο, σε πετρέλαιο με τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ξεχωριστά κάθε χώρα μέλος. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ε, και ένα άλλο σημείο, τελικό σημείο. Ε, ε συζήτησα με τον συνάδελφο μένα, αλλά γιατί κατ' ουσία ιδέα, εάν θέλουμε να πάμε σε μια ριζική μεταβολή του τομέα της κατανάλωσης της ενέργειας, ε, της παραγωγής των ΩΣΑ, αυτό δεν είναι ένα θέμα παρουσίασης. Γιατί δεν κινούμεθα σε μια ανάλυση μόνο σε συνάρτηση με τις ε, τιμές σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τους άλλους ε, δείκτες ε, ε, ή του Ιώζεφ Στίγκλιτς, επί παραδείγματι, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη ρύθμιση αυτής της δημόσιας συζήτησης. Είδω λοιπόν κάποια, κάποιες ενδείξεις ως δική μου συμβολή στην συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Πλάτιτ Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην εισηγήτρια για τις, ε, τους για την εξαίρετη δουλειά. Κάποια ζητήματα που προκύπτουν για συζήτηση. Στο ζήτημα του μηχανισμού τιμολόγησης καταρχάς και οι επιπτώσεις, οι λόγοι μάλλον που επηρεάζουν τις τιμές των αγαθών, τιμές των ε, πρώτων υλών, των καυσίμων κτλ. Αυτά όμως δεν ορίζονται μόνο μέσα από ένα μηχανισμό. Μπορούμε και με την ομοθεσία να ρυθμίσουμε τις τιμές. Και όπως και με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση αποδεικνύεται, πιστεύω, ότι η αγορά μόνη της δεν αρκεί για να ρυθμίσει τις αγορές. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να σπρώξουμε τις αγορές προς τη σωστή ρύθμιση των επιπέδων είτε επηρεάζοντα ε, με την εισαγωγή του μηχανισμού για την ε, σύλληψη και αποθήκευση άνθρακα, παραδείγματι. Και έτσι θα ήταν πιο ευχερή η επιτεύξη του στόχου για το διοξείδιο του άνθρακα κτλ. Και νομίζω ότι μπορούσαμε να κοιτάξουμε τα περιβαλλοντικά ε, ζητήματα πιο ουσιαστικά. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε και ανώτατα όρια στη χρήση των φυσικών πόρων ή των πρώτων υλών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην είναι τόσο αδύναμες σε σχέση με τη Ρωσία, την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εισαγωγές πρώτων υλών από εκεί. Επίσης για τον προϋπολογισμό και τις επιδοτήσεις έχουμε ένα τεράστιο σύστημα επιδοτήσεων για τον άνθρακα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Επιχορηγούμε το τετραπλάσιο από αυτό που περιμένουμε να εξασφαλίσουμε από το σύστημα των ε, τη εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών. Ε, α σταματήσουμε λοιπόν. Α κοιτάξουμε στου εθνικό μα προπολογισμού, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, πού βρίσκονται αυτέ οι επιδοτήσει και τι καταργήσουμε, διότι είναι ε, για την καινοτομία τελικά. Και εάν ούτω ή άλλω πρέπει να δούμε την ε, χρήση ε, των φυσικών πόρων από τα κράτη-μέλη, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και εάν πρόκειται να επιβάλλουμε χορηγήσεις, να χορηγήσουμε μάλλον επιδοτήσεις, ας ε, τις ε, χορηγήσουμε εκεί που μπορούν να προαγάγουν την καινοτομία. Και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι δεν επαρκούν οι φυσικοί μας πόροι, δεν έχουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε. Άρα θα πρέπει τα χρήματα που διαθέτουμε να ενισχύουν τους υφιστάμενους πόρους χωρίς να τους εξαντλούν. Τι χρηματοδότησή μας Φερρυπίν. Ευρωπαϊκή ή εθνική, εάν την ε, αυξήσουμε στο 20-30% και τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το αφήσουμε να το καλύψει η ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη οικονομία. Αυτό θα ήταν μια λύση. Επίσης, στα όσα έχουμε να ε, συζητήσουμε και να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ΕΡΑ, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Καθήκον μας είναι να ξεφύγουμε από την κρίση αυτή αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών μας μέσων και των πόρων μας, μέσα από τους προϋπολογισμούς μας, μέσα από τη χρηματοδότηση και τις λύσεις που μπορούμε να προβλέψουμε, δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αλλαγή τροχιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω. Θα ήθελα να μιλήσω στον εισηγητή για κάποια πράγματα. Ε, από ό,τι γνωρίζω, το σύστημα των δημοπρασιών ποσοστώσεων ε, δεν ξεκίνησε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2012 θα ξεκινήσει το σύστημα των δημοπλασιών. Αυτό που έχει τεθεί επιτάπητος είναι το εμπόριο ποσοστώσεων μετά Κιώτο, το οποίο υφίσταται και εφαρμόζεται μεταξύ χωρών. Δεν είναι πολλές, αλλά γίνονται κάποιες συναλλαγές με αντισυμβαλόμενα μέλη χώρες. Ξέρω ότι υπήρξε μεταξύ Ουγγαρίας, Ιαπωνίας, Λετωνίας, Αυστρίας. Είναι συμφωνία η τιμή ε, και είναι αποτέλεσμα η τιμή των του εμπορίου ποσοστώσεων μετά το και Όταν μιλάμε για αλλαγή του συστήματος δημοπρασιών ανταλλαγής ρήπων, εγώ δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καθιερωθεί το παρόν σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 εγώ συμμετείχα σε αυτή τη συνάντηση και ξέρω ότι οκτώ χώρες πολέμησαν για το 10% των ποσοστών να δίνεται χωρίς δημοπρασία στις χώρες. Αν αρχίσαμε να, να πουλάμε τα πάντα μέσω δημοπρασίας, θα αλλάξει η φυστάμενη απόφαση μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2012 το σύστημα, εγώ δεν θα συμφωνούσα να αλλάξουμε το σύστημα ε, όταν δεν έχει ξεκινήσει καν να λειτουργεί το νέο σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, πώς μπορεί να ρυθμιστεί η τιμή. Κανονικά, σύμφωνα με το σύστημα, αυτή είναι μόνο η αρχική τιμή της δημοπρασίας και αν κάποιος άλλος έρθει να αγοράσει, να αγοράσει στι εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα αυξηθεί τιμή. Θα πρέπει οι κυβερνήσει να καθορίζουν την αρχική ελάχιστη τιμή, αλλά δεν θα είναι η τελική τιμή. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Να, δεν μπορούμε να λέμε ότι εμεί θα καθορίσουμε την τιμή. Καλύτερο θα ήταν να επιταχύνουμε το πώς θα λειτουργεί το υιοθετηθέν σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην το αλλάζουμε πριν καν ξεκινήσει να λειτουργεί στην πραγματικότητα κανονικά. Ο κύριος Έγκελ. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω δύο πράγματα να πω. Το πρώτο είναι ότι μας λένε πάντα με αποφασιστικότητα και πεποίθηση που δεν πάβει να με εκπλήσει ότι η οικονομία του μέλλοντος θα είναι η πράσινη. τα πράσινα στοιχεία της οικονομίας έχουν κάποια υπεραξία οικονομική, αλλά έχω μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα της πράσινης οικονομίας να αντικαταστήσει όλα που έχουμε. Εδώ είναι η ουσία, στο κάτω-κάτω της γραφής. Μπορεί να δημιουργηθούν αισθέσεις απασχόλησης στα πλαίσια τα πράσινα, να υπάρχουν νέες δραστηριότητες πράσινες δεν είμαι πεπισμένος όμως ότι αυτή η πράσινη διάσταση της οικονομίας μπορεί να αντικαταστήσει κατά σημαντικό ποσοστό την οικονομία που γνωρίζουμε σήμερα. Και διαρωτώ αν είναι σκόπιμο και σωστό να διατηνόμεθα ότι μπορούμε να μετακινηθούμε σε πράσινη λειτουργία της οικονομίας αν στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, σε κάποια μέρη της Ασίας, μάλιστα έχω σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο αυτές τις περιοχές του κόσμου μπορούμε να, τις, ε, να εφαρμόσουμε μάλλον αυτά τα μέτρα, να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα σε πολύ λογικό χρονικό διάστημα. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει πολύ, αλλά λίμωνο, μόνο σε φιλοσοφικό επίπεδο, διότι πολύ λίγοι θέλουν να μιλήσουν μαζί μου γι' αυτό. Ε, c'est la notion du au-delà τι θέλω να πω. Πέρα από το ΑΕΠ, το, θέμα της μηδενικής ποσοτικής ανάπτυξης και πώς μπορεί να ε, ζήσει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα κράτη-μέλη μας και σε όλη την Ευρώπη τα επίπεδα ανάπτυξη στο μέλλον δεν θα τα πετύχουμε, δεν θα τα έχουμε. Και αυτό θα έχει σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση, χρηματοδότηση αυτού. Και τίθεται το ερώτημα. Μια που δεν θα χρειάζεται η οικονομία πάντα μια μεγάλη ποσοτική ανάπτυξη για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες τις κοινωνικές Εκεί αυτό δεν το διερευνήσαμε επαρκώς. Κυρίως όταν θα έχουμε μπροστά μας ε, μικρή οικονομική ανάπτυξη ποσοτικά εδώ στην ε, Ευρώπη και αυτή τη μακρά διάρκεια μικρής αναπτύξεως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, τις, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας που θα δοκιμαστούν. Donc, je vraiment que ça... Θα ήθελα λοιπόν αυτή η πτυχή να παίξει ρόλο επιφανή μάλιστα στα συμπεράσματά μας όσον αφορά την περίοδο μετά την κρίση. Που μπορεί να κρατήσει αρκετά αυτή η περίοδος της κρίσης και η περίοδος μετά την κρίση. Thank you very much, Mr. Chairman, Ευχαριστώ πολύ Κύριο Φέκμαρκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ στην ιδέα για μια νέα γεωργική πολιτική και άλλα θέματα. Σε άλλα όμω δεν συμφωνώ τόσο πολύ. Όπω είπε και ο προλαλή σα. χρησιμοποίησε τον όρο μετά κρίση, post crisis. Δεν είμαστε μόνο στην περίοδο μετά την κρίση. Είμαστε σε μια, στο κατόφλι μιας νέας εποχής και πρέπει να προετοιμαστούμε. Ταυτόχρονα βγαίνουμε από μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο δηλαδή της τελευταίας 30 ετίας. Τεράστιες ανάπτυξης εντυπωσιακής. Επίσης εξελίξεων εντυπωσιακών παντού. Και αν τα έγραφα αυτό το είχαμε δει πριν από 30 χρόνια, πιστεύω θα λέγαμε ότι είναι εμπνευσμένο από τη λέσχη της Ρώμης που επεσήμανε την έλλειψη πρώτων υλών. Το πέρας της χρήσης του χαλκού, την ε, εμφάνιση νέων μορφών ενέργειας και ούτω καθεξής. Αυτή ήταν η ζωφερή εικόνα που επικρατούσε την εποχή εκείνη. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Γιατί Είδαμε την εισαγωγή των ημιαγωγών νέων πρώτων υλών. Είδαμε μια διαφορετική λογική στη λειτουργία μεγάλων τμήματων της οικονομίας, νέες πηγές ενέργειας και τα τελευταία 30 χρόνια πολλοί άνθρωποι στον κόσμο και το περιβάλλον γύρω από αυτούς έχει, έχουν παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη. Από ένα δισεκατομμύριο έχουμε φτάσει στα τέσσερα, πολύ γρήγορα, μια ταχύτατη αλλαγή ως προς τις συνθήκες και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και ως προς την, ε, τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον μας. Επίσης τώρα, στις ενεργειακές πηγές. Βλέπουμε τώρα κάποιες νέες ενεργειακές πηγές και ήδη κάποιες από αυτές που ψεζόμαστε ότι μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Η δε υπόθεση ότι θα αντιμετωπίσουμε σπανίδα πρώτων υλών ναι, μπορεί να διατυπωθεί όπως είχε διατυπωθεί και πριν από 30 χρόνια. Ή ο εισηγητής αναφέρεται σε έλλειψη γεών. Δεν είναι αλήθεια αυτό έχουμε τεράστιες εκτάσεις ανά τον κόσμο και δεν αναφέρομαι στην περιοχή του Αμαζονίου εκτάσεις οι οποίες δεν αξιοποιούνται γεωργικά και αν αξιοποιούνταν γεωργικά θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά στο ανθρώπινο είδος. Επίσης η βιοενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα. Και ταυτόχρονα θα διαπιστώναμε και μια αναζωογόνηση περιοχών του κόσμου που ε, αντιμετωπίζουν τεράστια φτώχεια ακόμη, όπως είναι παραδείγματι ορισμένα τμήματα της Αφρικανικής Υπήρου. Άρα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να κοιτάξουμε το χρονικό μας ορίζοντα με ένα διαφορετικό μάτι, με ένα διαφορετικό πρίσμα. Και γι' αυτό θα αναφέρω και αυτό που είπε κάποιος άλλος συνάδελφος τις, κάποια άλλη συνάδελφος, τις επιδοτήσεις που έχουμε σε υπερβολικό βαθμό και οι οποίες ελαχιστοποιούν τελικά την ανάπτυξη. Οι διάφορες προτάσεις για φόρους που ακούμε. Εάν θέλουμε να επενδύει ο κόσμος περισσότερο, αν θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, τι τις θέλουμε τις φορολογικές επιβαρύνσεις, τι θέλουμε να φορολογήσουμε τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Δηλαδή να είναι πιο ακριβές, λιγότερο κεφάλαιο να είναι διαθέσιμο στα φτωχότερα μέρη του κόσμου. Να σταματήσει η ανάπτυξη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν συμφωνώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω ακόμη έξι συναδέλφους εγγεγραμμένους. Να σας διαβάσω τα ονόματα, έτσι να είστε έτοιμοι. Βάιγκελ, Χιούμπνερ, Γιάκον Σάρι, Γκίγκολτ, Χουντής και Τόμας Μάν. Βάγγελ, παρακαλώ. Βάγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι με εντυπωσιάζει το πράσινο χρώμα αυτής της έκθεσης και βεβαίως θα ήθελα να εγκομιάσω τον εισηγητή για τη διάρθρωση αυτή, για τη δομή αυτής της έκθεσης, γιατί πραγματικά μας ε, δίνει αρκετές ε, δυνατότητες για τη χάραξη μιας πολιτικής στο πεδίο αυτό. Έχω δύο σημεία ε, ερωτήσεις να θέσω. Υπάρχει κάποια υποκρισία, πιστεύω, όταν μιλάμε για τις ενεργειακές πηγές χωρίς να αναφέρουμε την ατομική ενέργεια. Πιστεύω ότι όλοι είμαστε εθισμένοι στις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει μια άτυπη, ένα άτυπη συμφωνίας να μην φύγουμε πλέον αυτό το θέμα ενώ πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σοβαρό θέμα των μελλοντικών ενεργειακών πηγών για πολλές χώρες. Η δική μου χώρα, για παράδειγμα, έχει ένα τρίτο της ενέργειας, ένα τρίτο της ενέργειας από ε, ατομικό, εργοστάσιο παραγωγής ατομικής ενέργειας το μόνο που υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε, να έχουμε την τόλμη να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να το θίξουμε. Το δεύτερο ερώτημα τώρα. Εγώ θα έδινα περισσότερη έμφαση στο, στο στο θέμα της έλλειψης ε, της ύδατος, υδάτινων πόρων. Γιατί μπορούμε να συζητούμε για το πού μπορούμε να βρούμε γη ή άλλες ε, πρώτες ύλε και να αναπτύξουμε νέες. Αλλά η δάτινη πόρη είναι γνωστή μόνο σε μία μορφή. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ, ότι σπανίζει το νερό όχι μόνο για την Αφρική, αλλά και για μεγάλα τμήματα της Ασιατικής Υπήρου ήδη Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να πούμε κάπως περισσότερα πράγματα για το θέμα των υδάτινων πόρων. Ευχαριστώ. Η Ντονάτα Χίμπνερ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που ότι εδώ υπάρχουν δύο εύλογα επιχειρήματα που θεωρώ ότι είναι πιστικά. Το ένα σχετίζεται με το ότι όλοι επιθυμούμε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας. Και το δεύτερο, ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας ε, σφαιρικά για μια πλήρη είσοδο στην ε, παγκόσμια οικονομία και στις ε, παγκόσμιες αγορές των δύο ή τριών παραπάνω δισεκατομμυρίων καταναλωτών τα επόμενα χρόνια. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο αποσιάζει από τη δική μας προσέγγιση σε αυτή τη, στο πλαίσιο της συζήτησης. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το Ότι η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη έχει πολύ, σημαντικές, πολύ ασυμμετρική παρουσία ε, ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή δεν έχουμε την ίδια εξέλιξη των κλιματικών αλλαγών. και αναλόγως τη μάχη θα τη χάσουμε στην Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να λησμονούμε ούτε την ξηρασία, ούτε τις πλημμύρες, ούτε τη διάβρωση των ακτών μας, ούτε όλα τα προβλήματα που βλέπουμε καθημερινά. Υπάρχει δε υψηλότερο κόστος και λόγω των τιμών ε, του άνθρακα και άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές ε, τις διαφορετικές παραμέτρους, ότι είναι ασυμμετρικές οι συνέπειες, ότι είναι ασυμμετρικές και οι ικανότητες ανταπόκρισης σε αυτές τις συνέπειες, και άρα μπορεί οι κλιματικές αλλαγές ε, να εντείνουν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, στην, ε, τα, την, την πρόοδο ή την ανάπτυξη μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποκλήσεις δηλαδή στην ανάπτυξη. Και βεβαίω οι τοπικέ αρχέ έχουν ευθύνη στην Ευρώπη, αλλά έχουν και διαφορετικέ αρμοδιότητε ανάλογα με τα πολιτικά συστήματα. Όταν κοιτάμε λοιπόν εν γέννη τη δομή του δημόσιου τομέα και του τρόπου λήψη αποφάσεων, εν γέννη τι επιλογέ στην Ευρώπη γενικά, τις καθημερινές επιλογές που θα ε, λάβει μια δημοτική αρχή, βλέπουμε ότι ε, τοποθετούνται στην... είναι οι αιτίε των ε, περαιτέρω εξελίξεων. Το αν θα υπάρχουν επαρκείς δηλαδή δημόσιες μεταφορές, το, αν θα είναι καθαρές οι μεταφορές, το αν θα μπορέσει ο κόσμος να μειώσει τη χρήση των αυτοκινήτων. Ο, κάθε επιλογή μιας δημοτικής αρχής έχει σχέση με την εξέλιξη των κλιματικών αλλαγών. Το τοπικό επίπεδο δηλαδή έχει τεράστια σημασία και ιδιαίτερα στην, στην, ε, ε, στον εντοπισμό των αιτιών των κλιματικών αλλαγών. Εάν λοιπόν δεν έχουμε επαρκείς προϋπολογισμούς με τις κατάλληλες προτεραιότητες, όσο καλά και είναι τα νομικά πλαίσια που εισάγουμε, δεν θα είναι αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Mm. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε για άλλη μια φορά και πιο αργά με κριτήριο νομίζω το εάν μπορεί να μας προσφέρει μία ενόραση για το μέλλον και να προβλέψει ενδεχομένως ε, κάποια νέα κρίση. Είπε ο κύριος Χόικμαρκ ότι έχουμε σε θέσή μας επαρκείς γεωργικές εκτάσεις. Έστω. Γιατί όμως μέχρι τώρα τα, τα πλούσια αραβικά κράτη αγοράζουν γη από τη Ρωσία. Οι, οι Φιλανδοί γιατί αγοράζουν γη από τη Ρωσία. Γιατί να σας πω. Διότι η γη είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας και μπορεί να οδηγήσει και σε οικονομικές φούσκες, απουνόφουσκες. Έτσι λοιπόν, μια και συζητούμε τις κρίσεις, δεν πρέπει να λησμονούμε και αυτό το παράγοντα. Την κερδοσκοπία επί των γεών. Για δε την πράσινη απόχρωση του εγγράφου. Ναι, είναι πολύ σημαντική η πτυχή αυτή. Αλλά δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο στα όσα έχουμε μέχρι τώρα κάνει μπορούμε να ακολουθήσουμε τις παλές μεθόδους. Πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να δούμε τι έχει να μας προσφέρει το μέλλον. Οι νέες τεχνολογίες. Πώς πριν από 20 χρόνια Φερρυπίν η χαρτοβιομηχανία μετατράπει σε μια ε, βιομηχανία high-tech υψηλής τεχνολογίας και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Ίσως λοιπόν θα ήταν ε, δυνατόν να δώσουν συγκεκριμένες ιδέες για το τι μπορεί να φέρει και για το βιομηχανικό κλάδο η πράσινη ανάπτυξη. Αυτή θα ήταν μια πιο ευφυής ενεργειακή πολιτική. Μια πολιτική και για τα οχήματα, οράματα γενικά που χρειαζόμαστε. Για δε το ηφαίστειο της Ισλανδίας, η έκρηξή του ήταν φυσικά, είχε καταστροφικές συνέπειες, αποτελούσε ταυτόχρονα και ένα μήνυμα, ε, να μια ένδειξη ότι τα πάντα μπορεί να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και θα πρέπει στην Ευρώπη πια να σοβαρευτούμε εντό εισαγωγικών, να κοιτάξουμε τα πράγματα με όριμο και σοβαρό τρόπο και να ξεκινήσουμε μια νέα αναγέννηση. να μην δαπανούμε αυτά που δεν έχουμε, να μην χάρουμε τις προοπτικές του μέλλοντος. Η πράσινη αυτή διάσταση, η προοπτική αυτή για το μέλλον πρέπει να γίνει πιο σαφής. Μέσα στο κείμενο πρέπει να πούμε πιο ξεκάθαρα το τι έχουμε να προτείνουμε. Ευχαριστώ. <clears throat> Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι κρίσιμη σημασία. Πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πετύχουμε το να καταλήξουμε σε μια έκθεση που είναι η βασική ιδέα δημιουργίας Επιτροπής της Κρίσης. Μια έκθεση που πραγματικά θα αντιμετωπίζει αυτή τη βαθιά κρίση και θα πετύχουμε ταυτόχρονα και μια νέα σύγκληση. Αν καταφέρουμε να γεφυρώσουμε το παραδοσιακό χάσμα που βλέπουμε στις διάφορες νομοθετικές επιτροπές, χάσμα μεταξύ συμφερόντων της οικονομίας από τη μία πλευρά και των συμφερόντων του πλανήτη από την άλλη πλευρά, αν καταφέρουμε να γεφυρώσουμε λοιπόν αυτό το χάσμα και αν θέσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο την οικονομική κρίση, το οικονομικό πλαίσιο τεθεί σωστά και λάβουμε υπόψη και τις κοινωνικές έντασεις, αν τα κάνουμε όλα αυτά, έχουμε μεγάλε πιθανότητε να πετύχουμε ευρεία συνένεση μεταξύ των διαφόρων ομάδων του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικότατο να συζητηθεί σοβαρά το θέμα, ή μάλλον τα θέματα. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια από τα σημεία που εθίγησαν ο κ. Χόκμαρκ. Κύριε Χόκμαρκ, είναι σημαντικό να σας πω το εξή: Αυτή η έκθεση πριν από 30 χρόνια δεν θα μπορούσε να συγγραφεί από κανένα του πράσινου κινήματος. Έχει υποθέσεις και συμπεράσματα που διαφέρουν κατά πολύ από την παραδοσιακή θάση του πράσινου κινήματος, το παρελθόντος. Ε. Το τονίζω αυτό διότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η έκθεση στα μέσα που αναφέρει για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι αγορές παίζουν σημαντικό ρόλο τελικά, θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να επιφέρουν την αλλαγή. Και παίρνει μια θέση έκθεση στο δογματικό θέμα της ανάπτυξης για το πράσινο κίνημα δογματικό. δεν κρίνει αν είναι καλό ή κακό η ανάπτυξη. Στο παρελθόν το πράσινο κίνημα έλεγε δεν θέλουμε, μεγάλη, δεν θέλουμε άλλη ανάπτυξη. Εδώ η έκθεση λέει ότι το ΑΕΠ δεν είναι το σωστό μέτρο προσμέτρησης της ευμάρειας και της ευζοίας. Και λέει η έκθεση ότι πρέπει να μειώσουμε το βάρος που θέτουμε στον πλανήτη. Να μην καταστρέψουμε τον πλανήτη. Αλλά πόσο ΑΕΠ συνάδει αυτό τον στόχο ε, δεν το λέει η έκθεση και έχει τους λόγους της. Προσπαθούμε μέσω της εκθέσεως να κάνουμε μια πρόταση. Σας ευχαριστώ για αυτό. Πρόταση που ταιριάζει με το στόχο μας. Στόχος μας είναι η προστασία του πλανήτη. Και ταυτόχρονα γίνεται αποδεκτή και μια θέση που δεν είναι παραδοσιακά πράσινη. Άρα είναι θέμα προς συζήτηση. Αν αμφισβητούμε το ρόλο της αναπτύξεως του ΑΕΠ που θεωρείται κρίσιμο στόχος, να σκεφτούμε μήπως μπορούμε να βρούμε μια θέση επί της οποίας να συμφωνήσουμε. Ότι δεν είναι αυτός σκοπός να βρούμε άλλο τρόπο να να κινηθούμε για να πετύχουμε καλό επίπεδο διαβίωσης πέρα του ΑΕΠ και να χρησιμοποιούμε σωστά τους πόρους του πλανήτη. Στο ερώτημα ποιο είναι το ενδεχόμενο μέγεθος της πράσινης οικονομίας. Άλλο κρίσιμο σημείο. Που πιστεύω ότι είναι σημαντικό για να γεφυρώσουμε κάποια ενδεχόμενα χάσματα. Η πράσινη οικονομία ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους. Μερικοί λένε έχουμε τι εγκαταστάσει με άνθρακα, πυρηνικέ μονάδε παραγωγή, έχουμε τα αυτοκίνητα που ρηπαίνουν, παραδοσιακή κατανάλωση κρέατος με παραδοσιακό τρόπο γεωργίας. Και τώρα έχουμε νέα πηγή ανάπτυξη. Πάνω σε αυτά προσθέτουμε και ωραία ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τους πράσινους, κάποια χορτοφαγικά πιάτα για τους πρασίνους. Προσθέτουμε και ανανεώσιμους πόρους Χημική βιομηχανία βασίζεται σε όμω πόρου. Πολύ ωραία. Άλλη μια πηγή ανάπτυξη προσθέτουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη βάση, δεν μπορούμε να πετύχουμε σύγκληση με αυτή την προσέγγιση, γιατί ο πλανήτη πάλι θα καταστραφεί. Από τι παλιέ μορφέ τι βιομηχανικέ. Άρα δεν θέλουμε αυτό. Τι θέλουμε. Οι παλιέ καταστροφικέ μορφέ βιομηχανία και κατανάλωση να αντικατασταθούν. Να αντικατασταθούν από ένα είδο κατανάλωση που να είναι φιλική προς τον πλανήτη και που προστατεύει και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων. Και αυτό θα μπορούσε να ταιριάζει και με το, την καθαρή αύξηση του ΑΕΠ και την καθαρή αύξηση της απασχόλησης. Μπορεί να ισχύσει αυτό και αν συγκλίνουμε. Τέλος. Ακροθυγός. Η λέσχη της Ρώμης έκανε λάθος το είπατε κι εσείς, το είπαν και άλλοι, ότι είναι, αν ακολουθήσουμε την πορεία θα, σταματήσουν, θα τελειώσουν οι πρώτες ύλες. Είναι δυνατόν η ανθρώπινη δημιουργικότητα να βρει αντικατάσταση για σπάνιδα σε κάποια είδη, ε, σε κάποια προϊόντα. Αλλά είναι ανοιχτό το στοίχημα. Δεν ξέρουμε αν ισχύει. Δεν ξέρουμε αν από τους σπάνιους πόρους θα αντικατασταθούν αποτελεσματικά από κάτι άλλο. στις τιμές το βλέπουμε ότι σε κάποιες αγορές υπάρχει δυσκολία και αυτό θα είναι οικονομικό πρόβλημα. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μεγάλη σημαντική φορείς και βασικά ερευνικά ιδρύματα το εξετάζουν το θέμα του τέλους των πόρων. Αυτό είναι τεράστιο κίνδυνο για την οικονομία εάν για βασικούς πόρους, για πρώτες ύλες δεν υπάρχει καλό υποκατάστατο. Σαν οικονομολόγος λοιπόν, κατευθυνόμενος από την αρχή της πρόληψης, σαν οικονομο... θα πρέπει, λέγω, ότι θα πρέπει να είμαστε αποδοτικοί, αποτελεσματικοί όσον αφορά την χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ λέω ότι στη συζήτησή μας θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα και να προσπαθήσουμε όλοι να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Ποιο χάσμα μεταξύ των διαφόρων παραδοσιακών ιδεολογιών ε, για να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάτι που θα το παρουσιάσουμε σαν Επιτροπή και να πούμε ότι να βρήκαμε κάτι που είναι πιο πέρα από τις παραδοσιακές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την σοβαρή δουλειά και για το κείμενο που έχει κάνει, διότι εκτός των άλλων μας θυμίζει δύο πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Το πρώτο ότι η κρίση που βιώνουμε δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, δεν είναι μόνο κρίση χρηματοπιστωτική, είναι και κρίση περιβάλλοντος, όπως είναι και κρίση ενεργειακή και κρίση διατροφική. Και επομένω με, μια, με αυτή την ευρύτερη θέαση πρέπει να, δούμε, να βλέπουμε τα μέτρα εξόδου από την κρίση και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και το δεύτερο είναι ότι μας θυμίζει ή τουλάχιστον υπογραμμίζει ότι ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο ΑΕΠ, ότι η ανάπτυξη και η πραγματική ευημερία είναι πέρα πολλές φορές από τους αριθμούς και τα νούμερα. Μου θύμισε μια έκφραση που λέμε στην Ελλάδα ότι καμιά φορά μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Για αυτές τις δύο βασικές θεάσεις της κατάστασης με βρίσκει σύμφωνη η έκθεση όμως εδώ μετέχοντας σε μια συζήτηση και νίκη της οποίας έκανε και ένας συνάδελφος πριν <clears throat> είναι η πυρηνική ενέργεια μέσα στις εναλλακτικές προτάσεις που αναζητούμε αυτή την περίοδο. Βλέπω ότι επανέρχεται το θέμα αυτό. Είχε πράγματι μπει στο περιθώριο μετά από τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί με το Τσέρνομπιλ και αλλού και εμφανίζεται ως μια εύκολη λύση οικονομική, καθαρή, όλα αυτά εντό εισαγωγικών. Νομίζω ότι είναι λάθος η προσέγγιση, δεν συμφωνώ βεβαίω. Είναι μια προσέγγιση που λέει έχουμε πρόβλημα διατροφικό, έχουμε διατροφική κρίση, πάμε στα μεταλλαγμένα. Έχουμε πρόβλημα περιβάλλοντος, πρόβλημα ενεργειακό, πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά βλέπω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί ευρύτερα το επόμενο διάστημα και επομένως νομίζω ότι πρέπει να μπει και στη δική μας προβληματική ε, και σε πιο αναλυτική και διεξοδική συζήτηση σε σχέση βεβαίως με την επιπτώ, τις επιπτώσεις της και στα, ε, στην γενικότερη οικονομική προοπτική. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε δύο συγκεκριμένα θέματα της έκθεσης και με αυτά να τελειώσω. Ε, το πρώτο έχει να κάνει με το σύστημα εμπορίας ρήπων. Εδώ, να μου επιτρέψετε ε, να διατυπώσω πολλά ερωτηματικά και πολλές ενστάσεις δηλαδή όσο αφορά την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος και βεβαίως με τον τρόπο που γίνεται. Εδώ τώρα τι κάναμε, αντί να γίνει πιο αυστηρή, πιο απαιτητική η πολιτική, οι πολιτικές, τα μέτρα για τον βεριοσμό των ρήπων, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές ε, ε, χώρες, δημιουργήθηκε μια νέα αγορά όπου πρωταγωνιστούν οι ήδη οι κερδοσκόποι και συνήθεις ύποπτοι των ε, διεθνών χρηματαγορών. Με πολύ αμφίβολο το αποτέλεσμα όσο αφορά τη μείωση των ρήπων. Ε, αναρωτιέμαι, ίσως στην, ε, στο δευτερολογία του εισηγητής, ε, πώς το βλέπει αυτό το... Ασκεί, κριτική στο σύστημα εμπορίας, αλλά τελικά θα αποδεχθούμε αυτή τη λογική της εμπορευματοποίησης, της διαδικασίας ελέγχου, της κλιματικής αλλαγής. Θα το κάνουμε εμπορευματικό μέγεθος και αυτό. Εκείνη η ενστάση θα ήθελα κάτι παραπάνω από τον εισηγητή. Και το δεύτερο, σε σχέση με τα μέτρα και τις χρηματοδοτήσεις ε, για τη μετάβαση, την τεχνολογική μετάβαση των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων, ε, γιατί πρέπει το βάρος και πάλι να πέσει σε διορθωτικά ταμεία, σε κρατικούς προϋπολογισμούς και όχι να υπομιστούν μεγαλύτερο βάρος αυτές οι βιομηχανίες και αυτές οι επιχειρήσεις που τόσο καιρό ρήπαιναν και εκμεταλλεύονταν αυτή την ε, μονοπωλιακή τους θέση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Τόμας Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον συνάδελφο κύριο Γκίγκολ και άλλου ότι το θέμα τη προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των πρασίνων, αλλά και άλλε χώρε μέλη, άλλε πολιτικέ ομάδε έχουν εντάξει το θέμα αυτό και αυτό είναι σημαντικό. Ε, και θέτουμε κάποιε προποθέσει κι εμεί, όπω και οι πράσινοι για το περιβάλλον, αλλά η ανάγκη να αναλάβουμε ευθύνη, να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, να συζητούμε για μια βιώσιμη πολιτική, νομίζω και να αγωνιζόμεθα για αυτήν, νομίζω ότι αυτό ισχύει για πολλές πολιτικές ομάδε. Βεβαίω υπάρχουν ορισμένε θέσει για τι οποίε μπορούμε να συζητήσουμε τι είναι εφικτό σήμερα και τι είναι εφικτό μελλοντικά. Όταν λέμε ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο, αυτό κάτι σημαίνει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε την ε, χρηματοπιστωτική κρίση ε, και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους άλλους τομείς. Υπόθηκε ότι υπάρχει η διατροφική πολιτική, το θέμα της πολιτικής των συγκοινωνιών, της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου δεν έχουμε μεν ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά είναι επίσης ένα σημαντικό τομέα. Αλλά δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα σε αυτή την έκθεση. Νομίζω θα πρέπει κάπου να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Η Περβάνς Περές δεν μπορεί να εντάξει τα πάντα σε μια κρίση όπου επιθυμούν να έχουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ωστόσο, ορισμένα σημεία θεωρώ ότι είναι ορθά. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων. Ο ε, κ. Ρότιγκεν θα εκπληρώσει πολύ καλά τις, τα καθήκοντά του νομίζω. Από την άλλη θα πρέπει να κινήσουμε ε, κάποια, να εργοποιήσουμε κάποια κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ε, πολιτικής ε, μεταβολής, της κλιματικής μεταβολής, συγγνώμη. Στη Γερμανία έχουν ήδη επιτευθεί κάποια πράγματα Θεωρώ παρόλα αυτά ορθό οι χώρες μέλη να χαράξουν το δικό τους δρόμο και να μην επιληθεί το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι θα υποφεληθούμε από σωστά μέτρα, γιατί και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό ερέθισμα. Όσον αφορά το ζήτημα του φόρου Τόμπιν, εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Γιατί εάν επιβληθούν τέτοιου είδου φόροι, θα πρέπει να επιβληθούν και σε έναν σημαντικό ενεργειακά τομέα, όχι μόνο για να κλείσουν οι τρύπε του προπολογισμού. Όσον αφορά τα διορθωτικά ταμεία, εδώ αναφέρθηκε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντική η ύπαρξή του γιατί θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα αναπροσανατολισμού επαγγελματικού των εργαζόμενων. Μια δέσμη μέτρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και όχι μόνο να επενδύουμε στους πράσινους ε, τομείς και μόνο. Αυτό αφορά ε, πάρα πολλούς άλλους τομείς. Εμείς στην Επιτροπή Απασχόλησης είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα και χαίρομαι ε, που μπορούμε επιτέλους να πούμε ότι η Ευρώπη δεν βοηθάει μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικές οι προσεγγίσεις αυτές της έκθεσης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν κατάλληλα οι σημαντικές προτεραιότητες και η υπερβάνωση θα πρέπει να αναλάβει αυτό το έργο, να δώσει τη σωστή έμφαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ δεν διεκδικώ αποκλειστικά τα πράσινα θέματα και αυτό συνείδητα το λέω προς τους Βρετανούς συναδέλφους. Δεν πρόκειται εδώ για μια έκθεση της Λέσχης της Ρώμης. Η Λέσχη της Ρώμης ε, ε, κατάληξε μια εντελώς διαφορετική έκθεση. Αν τη δείτε είναι γεμάτη από καινοτόμα στοιχεία, προς αγγλισμό, προς την αγορά, προς εντελώς ε, καινούργια πράγματα που θεωρώ ότι συνιστούν ένα νέο κίνημα, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος κ. Γκίγκολτ. Γιατί εδώ κοιτάμε για το προγραμματισμό νέων συνασπισμών για τη δημιουργία μια νέα μελλοντική οικονομία. Εγώ προέρχομαι μένα από το Πράσινο Κόμμα, αλλά αυτή είναι ίσω μια ε, σύμπτωση, αν θέλετε. Δεν είναι ένα καθαρά πράσινο έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο που αφορά ε, τον προσανατολισμό προ μια νέα οικονομία και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινή βάση, πράγμα το οποίο άλλωστε εξέφρασαν πολλοί συνάδελφοι. Μπορούμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό. Ορισμένοι από εσά ε, εξεπλάγησαν που ήταν μια, ένα πράσινο έγγραφο. Αλλά δεν είμαι πράσινος όπως σας είπα. Τώρα, αν επανέλθουμε στη, λέσχη της ε, Ρώμης. Ο, συντα... ο συγγραφέας της λέσχης της ε, Ρώμης ε, ασχολείται με το θέμα αυτό και καταλήγει ότι για τα ενεργειακά θέματα η προβλέψεις αφορούν ορισμένες, ε, ορισμένους τόχους. Εμείς δείχνουμε ότι αν εξετάσουμε την ανάπτυξη του, το ζήτημα του πετρελαίου, ε, βρίσκουμε ότι ίσως ε, είχαν δίκιο σε κάποια θέματα, στο θέμα της ενέργειας. Σε ορισμένα θέματα είχαν δίκιο, σε άλλα όχι. Ε, μπορεί κανείς να αξιοποιήσει κάποια από τα συμπεράσματά τους. Αλλά ε, βεβαίω τώρα είμαστε πολύ μακριά. Αυτές οι εκθέσεις γράφτηκαν τη δεκαετία του 70. Τώρα, όσον αφορά την ε, προοπτική του χρόνου, συμφωνώ για τα όσα είπατε, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αν αφήσουμε μόνο στη ρύθμιση των αγορών τη δυνατότητα ανάπτυξη νέων βιώσιμων πράσινων οικονομιών και μία αποτελεσματική οικονομίας, το ζήτημα είναι ότι οι αγορές αποκρίνονται ε, πολύ αργά, με πιο βραδείς ρυθμούς. Η κοινοτομία βεβαίως μπορεί να επιλύσει πολλά πράγματα, αλλά θα εισαχθεί εγκαίρως. Λόγω ακριβώς της ε, πίεσης χρόνου νομίζω θα πρέπει να υπάρξει χάραξη πολιτικών για να προλάβουμε, γιατί αν περιμένουμε έως ότου υπάρξουν ορθά ε, ε, κίνητρα μέσω της αγοράς, θα, θα στοχίσουμε. Γι' αυτό ακριβώς έγραψα αυτή την έκθεση. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα της γης, γιατί και εδώ μπορούμε να έχουμε πάσης φύσεως ενδιαφέρουσες ε, συζητήσει. συζητήσεις. Εγώ κάνω μια έρευνα σε αυτό το χώρο πριν γίνω βουλευτής και αν δούμε τι γίνεται στη Γεωργία, 40% της χρήσης ε, γης ε, καλύπτεται από τη Γεωργία. 20% Μιλάμε βεβαίως και για εκτάσεις τούντρας, ερήμους κλπ. Αν δούμε και τη δασική κάλυψη, ε, η διαθεσιμότητα της αρωτρέας ε, γης δεν είναι τεράστια. Ορισμένες ε, χώρες, όπως υπόθηκε, αγοράζουν γη από αναπτυσσόμενες χώρες γιατί ακριβώς ε, συνειδητοποιούν αυτό το πρόβλημα. Το μείζον θέμα είναι λοιπόν πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα και πάλι ένα ζήτημα καινοτομία. Αλλά αυτό στο οποίο στοχεύω είναι ότι αν ε, απλώς βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της γης ε, μέσω ε, λιπασμάτων, η τιμή των λιπασμάτων συνδέεται με την τιμή του πετρελαίου. Άρα επιφέρει κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το ζήτημα της καινοτομία και της αξιοποίησης των πόρων. Ορισμένοι λένε πώς ε, μπορείτε να είστε τόσο σίγουρος ε, ότι η πράσινη οικονομία είναι μια υπόσχεση για το μέλλον. Μπορούμε να το διατυπώσουμε διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι μελλοντικά θα πρέπει να, πράγματι να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους. Η Κίνα είναι ηγέτη στην ηλιακή ενέργεια, θα γίνει ηγέτιδα δύναμη και στην ηλιακή ενέργεια, στην αιωλική ενέργεια. Ε, θέλουμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό τους παράδειγμα ή να ακολουθήσουμε από πίσω, θέλουμε να είμαστε και εμείς ε, σε, στην πρωτοπορία αυτής της νέας οικονομίας. Ε, θα είμαστε στην προμετωπίδα ή θα στερούμε πίσω μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα προτιμούσα να δώσω περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά είχα έναν περιορισμό στην έκθεσή μου σελίδων λέμε δώστε μας διαφανείς προβλέψιμες πολιτικές για να μπορέσουμε να κατατείνουμε προς κάποιους στόχους. Εσείς που χαράζετε την πολιτική, δώστε μας διαφανείς πολιτικές. Αυτό είναι το ζήτημα, το ζητούμενο. Γι' αυτό λοιπόν διατυπώνω και εγώ αυτό το αίτημα. Βεβαίω είχα έναν περιορισμό, όπω είπα, έκταση στην έκθεσή μου και δεν μπόρεσα ίσω να το πόσο πιο ξεκάθαρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά δεν πρόκειται εδώ για ένα πράσινο χόμπι. Είναι για το μέλλον όλων μα. Ευχαριστώ πολύ. Θα, Θα περάσουμε τώρα στο τέλο του πρώτου τμήματο. Και τώρα να δούμε το έγγραφο εργασία υπαριθμών 7, το επόμενο σημείο, Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Διεθνή Νομισματική Πολιτική και Αντιμετώπιση των Παγκόσμιων Ανισορροπιών. συμπεριλαμβανόμένων του ζητήματο των φορολογικών παραδείσων. Ο Κ. Σουίνμπορν είναι ο θεματικό συντονιστή. Τον καλό να μα κάνει την παρουσίαση του θέματο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι θα είδατε κι εσείς ότι ήταν δύσκολο, πως και για τους συναδέλφους, να περιορίσω το τεράστιο αυτό θέμα στις 7 σελίδες. Για το κάθε ένα από τα τρία ε, θέματα θα μπορούσα να είχα γράψει βιβλίο ολόκληρο. Και για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχει η πιο εκτενής μορφή πέραν των 7 σελίδων. Δηλαδή πολύ ευχαρίστως να σας δώσω επιπλέον υλικό. Να διαβάζετε τη νύχτα για τη μυθιστόρημα. Έχουμε λοιπόν ε, προβλήματα με τις ανισορροπίες, την, ε, τα, την, την κρίση τη διακυβέρνηση, την ρυθμιστική διακυβέρνηση, τη μεσηματική πολιτική και σκοπός της έκθεσης είναι να εξετάσει επιπτώσει αυτών των παραγόντων και να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματο εναντί ενός μελλοντικού κλειδονισμού αντίστοιχου μεγέθου. Αλλά αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι περιορίζονται μόνο σε αυτού του τρει παράγοντε. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην κατάσταση. Τη χρηματοπιστωτική πολιτική επίσης τις δομές των ε, τραπεζών, την υπερβολική εξάρτηση από μαθηματικά μοντέλα κινδύνου με συνέπειες πολύ σημαντικές. Επίσης βλέπουμε το τον συνδυασμό αυτών των ε, ελλείψεων ως κύριο παράγοντα της αποτυχίας του συστήματος. Η κρίση λοιπόν το 2007 με 2009 στις ε, ε, χορηγίες των, χορηγίες των δανείων ήταν ε, η πρώτη ένδειξη της κρίσης και ίσως μπορούμε να κοιτάξουμε ιστορικά την κρίση. Όταν το 1995 μπήκε η Κίνα στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ε, ένα σημαντικό βήμα προς την παγκοσμιοποίηση. Είχε βέβαια μεγάλο πλεόνασμα μέχρι τη δεκαετία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 η Κίνα και οι μεγαλύτερες οικονομίες είχαν περάσει στον βραχυπρόθεσμο δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη στόχο της ισοτιμίας με ένα κάνιστρο ε, προϊόντων και, και υπηρεσιών. Ε, ως νέο σύστημα, ενώ στο παρελθόν, στη δεκαετία του 80, οι Ηνωμένε Πολιτείε Τετέρωση για να καταγράφουν την ανάπτυξη είχαν ε, ε, ένα σύστημα νομισματικό χρησιμοποίηση. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και προς το τέλος στην κρίση των ασιατικών κρατών, το 98 στην, στην κρίση της διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ένα πρώτο σήμα κινδύνου αν θέλετε της σημερινής κρίσης, και ένδειξη των όσων θα μπορούσαμε να περιμένουμε, δηλαδή υψηλό επίπεδο ανεργίας, αρνητικές συνθήκες στην αγορά και συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση του συστήματος. Το 1999 ε, εισήχθη το ευρώ με ορισμένες χώρες, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία και ε, Πορτογαλία και Ιταλία ιδιαίτερως που δεν είχαν επαρκώς ε, φτάσει στους όρους της συνθήκης του Μαστρίχτ και που είχαν προβλήματα και λόγω των ανισορροπιών στις εσωτερικές τους οικονομίες. Και άλλα στοιχεία βέβαια εντάξει στο πλαίσιο αυτή τη κρίση, αλλά αν κοιτάξουμε τι παγκόσμιε ανισορροπίε, είναι σημαντικό να ορίσουμε τι εννοούμε ω ανισορροπία με την έκθεση αυτή, διότι σημαίνει ότι δεν έχουμε ε, η συμμετρία και ότι ξεφεύγουμε από την ισορροπία. Άρα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επικίνδυνες αρισορροπίες και ποιες είναι μάλλον ε, θετικές, οι καλοήθεις. Υπάρχουν λοιπόν ανισορροπίες σε όλες τις αγορές, τις αντισταθμίζουν όμως οι παράγοντες της αγοράς και μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα μετάβασης. Και αυτό καταγράφεται στα περισσότερα ε, μοντέλα τιμολόγησης και λειτουργίας της αγοράς. Υπάρχει παραδείγματι η υπερβολική εξάρτηση στις εξαγωγές ή τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές του ρωμανου Βασίλειο, εξαγωγές Γερμανία, Κίνα. Ε, άλλες ανισορροπίες μπορεί να υπάρχουν ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα ή τα πλεονάσματα που μπορεί επίσης να επηρεάσουν τις ανισορροπίες. Όμως αυτές δεν είναι ανεξάρτητες της κρίσεως. Μένα μπορεί όμως και να επηρεάσουν τη δυνατότητα μιας συγκεκριμένη χώρας να αντιδράσει στην κρίση. Η εξαίρεση νομίζω σε αυτά τα μοντέλα είναι η κατάσταση του ελλείμματος των ΗΠΑ και του πλεονάσματος της Κίνας και τα διαρκή πλεονάσματα των ε, πετρελαιοεξαγωγικών κρατών που έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, στα φαινόμενα των τελευταίων ετών. Άλλη μια μεγάλη κλίμακα ανισορροπία είναι αυτό το οποίο έχουμε δει από τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπου έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους ε, για διάσωση ορισμένων χαρών και θα μπορούσα να δώσω ε, κάποια παραδείγματα γιατί αυτές οι επενδυτικές τράπεζες έχουν συμβάλει στην ε, κρίση. Ότι δηλαδή σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και για πολλούς λόγους δεν υπήρχε δυνατότητα να προσαρμοστεί ε, η αγορά στις σύγχρονες ε, συνθήκες ένα μια δυνατότητα να προσφέρονται οι υπηρεσίες και τα αγαθά στους μεγαλύτερους ε, πελάτες ήταν περισσότερο ο στόχος ο οποίος οδήγησε στην προσπάθεια της διόγκωσης των επιχειρήσεων και έτσι μικρότερες επιχειρήσεις προσπαθούσαν μόνο να διόγκωθούν για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα πελατολόγια. Οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις προσπαθούσαν να βρουν μεγαλύτερα κομμάτια της αγοράς στη διάθεσή τους και έτσι είχαμε εκρηκτική ανάπτυξη και στον χώρο των χρηματοπιστωτικών παραγόντων που δεν υπήρχαν καν μερικά χρόνια πιο πριν. Όλοι οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ε, εξαπλώθηκαν κατά τρόπο εκρηκτικό και επιθετικό με τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα, χωρίς να είναι όμως αντιληπτός και ο κίνδυνος στον οποίο εμπλέκονταν. Και ναι, δεν μπορεί ίσω κανείς ε, να καταλαβαίνει κάθε είδους λεπτομέρεια των μαθηματικών αυτών μοντέλων, πλην όμως θα έπρεπε αυτοί οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να γνωρίζουν τι σημαίνει το τοξικό μείγμα χαμηλών ε, αποδόσεων υψηλού κινδύνου και αντί να ε, θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι ο κίνδυνος θα ήταν ε, ότι δεν θα μπορούσαν να μεγαλώσουν, να διακοδοθούν ακόμη περισσότερο, μάλλον ε, φοβόντουσαν ότι δεν θα, ε, ότι δεν, μάλλον θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να αποτύχουν. Ήταν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή που δεν θα μπορούσαν ποτέ να, να αποτύχουν. Ταυτόχρονα η αποταμίευση και ο δανεισμός, ενώ κανονικά σε, παγκόσμιο επίπεδο είναι σε ισορροπία, δηλαδή έχει μηδονικό υπόλοιπο, θα πρέπει να έχει και ένα, μια ισορροπία που όμως τα τελευταία, τελευταία δεκαετία ανατράπηκε τα τελευταία χρόνια στην Κίνα με το υψηλό πλεόνασμα και σιγά σιγά και στις πετρελαϊκές χώρες. με, εσφαλμένες, με συγκεκριμένες επιλογές μάλλον, Κίνα δηλαδή η οποία προήγε μάλλον τις εξαγωγές εις βάρος της εσωτερικής κατανάλωσης, με μια συγκεκριμένη φορολογική πολιτική, με ένα συγκεκριμένο σύστημα ε, ισοτιμιών, νομισματικών ισοτιμιών, με ζητήματα και ως προς την ιδιωτική περιουσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φορολογία μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών που οδήγησαν στις ε, συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε και τις επιπτώσεις τους στο παγκόσμιο εμπόριο. Αν και δεν νομίζω ότι ε, αν δεν αντιμετωπιστεί η εσωτερική κατανάλωση στην Κίνα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Φαίνεται ότι οι αρχές της Κίνας επέλεξαν αυτό το πρότυπο, θεωρώντας ότι έτσι έχουν περισσότερα να κερδίσουν, συμπιέσοντας δηλαδή την ιστορική τους κατανάλωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και να συζητήσουμε. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη ακόμη και στις ε, χώρες ε, παραγωγούς πετρελαίου, λόγω και της αύξησης ε, των τιμών του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, που έχουν χαμηλή κατανάλωση και γενικά χαμηλό κόστος ως προς την κοινωνική ασφάλιση και έτσι μπορούν να ενισχύσουν την αποταμίευση σε εσωτερικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας δε για τα νομισματικά τους αποθέματα το δολάριο, ε, ενθαρρύνουν την αποταμίευση σε δολάρια. Ναι, αυτή λοιπόν η ανισορροπία σχέση με τις ΗΠΑ ήταν καλοήθης για τις ΗΠΑ ε, για, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε την εξής εικόνα. Από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ε, είδαμε ελλείμματα στα τέλη της Προεδρίας του Μπούς. Χωρίς αύξηση των επιτοκίων, έτσι θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Αλλά επειδή εισέρεαν χρήματα από την Κίνα και από ξένους δανειστές, ε, επηρεάστηκαν αντίστροφα τα επιτόκια με αποτέλεσμα να ενισχυθούν και τα σπρέτς. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο και, και έχει την ε, μεγαλύτερη χρήση ως ε, γνώμονα στις συναλλαγές στο δολάριο. Η αγορά των ε, ακινήτων και ιδιαίτερα των κτηματικών ελληνικών ε, δανείων ε, στις ΗΠΑ επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο. Τα ποσοστά, τα επιτόκια που χορηγούνται για τα δάνεια επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Και στο χρηματοπιστωτικό τομέα ιδιαίτερος βλέπουμε και χαμηλότερες απαιτήσεις για το κεφάλαιο και Ε, συστήματα ενίσχυσης του κέρδους αναμετοχή, τα οποία ανατρέπουν ολόκληρο το παραδοσιακό σύστημα του χαρτοφυλακίου, των μετοχών δηλαδή. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι ένα φθηνό δάνειο, επειδή υπήρχε σχετική ευνοϊκή φορολογία, ε, θα μπορούσε να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τις μετοχές τους. Σε αυτό βλέπουμε ότι η φορολογία επηρέασε την κρίση, ενίσχυσε την κρίση δηλαδή, αλλά ε, η φορολογική παράδειση είχαν και αυτή κάποια επίπτωση. Εγώ προσπάθησα να κοιτάξω λίγο την αποταμίευση στους φορολογικούς καταλόγου, ε, παραδείσους, χωρίς όμως συγκεκριμένα αποτελέσματα πρέπει να πω. Με συγχωρείτε, η φωνή μου δεν ε, πάει πολύ καλά, έχω βραχνιάσει. Είναι ειδικέ οντότητε αυτή η φορολογική παράδοση. Είναι ουδέτερη φορολογικά. Στόχο έχουν να ενισχύσουν τις ε, ε, επενδύσεις και μπορεί να αναστέλλονται οι φορολογικέ υποχρεώσει, αλλά δεν απαφεύγονται τελείως. Άρα δεν είναι πιθανόν αυτέ οι φορολογικέ έδρε των οντοτήτων να ήταν κινητήρια δύναμη πίσω από τη σύστασή του και να μην δραμάτισαν κύριο ρόλο στο πρόβλημα που ανέκυψε. Η διαχείριση τώρα αυτής της κατάστασης ε, από τις μεγάλες, ε, τις κεντρικές τράπεζες παραδείγματι που διατήρησαν πολύ χαμηλά τα επιτόκια, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία ε, διαρκώς επέκριναν οι οικονομολόγοι της αγοράς, διότι δεν επέτρεπε την ανάπτυξη των ε, κερδών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζώνης του ευρώ, ορισμένες κυρίως από αυτές. Χρειάζεται λοιπόν μια πιο, προσ... πιο εστιασμένη προσέγγιση ως προς το ζήτημα των επιτοκίων και για να σταματήσω να διαβάζω το κείμενό μου θα προχωρήσω στο τελευταίο ζήτημα που έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση. Υπάρχει ένα κύριο ζήτημα, ένα ζήτημα ως προς την ε, εταιρική διακυβέρνηση αλλά και ως προς τα κράτη-μέλη και την παγκόσμια διακυβέρνηση. Θα πρέπει, πιστεύουμε, οι εκτός ε, ισολογισμού συναλλαγές από επιχειρήσεις και κράτη να καταργηθούν οι δυνατόν και με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση τα κράτη μόνα τους δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Υπάρχουν ε, παράγοντες, ε, ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ανεξάρτητα από τα μέτρα που λαμβάνονται στο αποτέλεσμα της κρίσης θα υπάρξουν και στο μέλλον οικονομικοί κλειδονισμοί. Το κράτο είναι ασφαλιστή έσχατη ανάγκη και επιμένω αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του περιθωρίου δημοσιονομικών ελιγμών. Και ναι, μπορεί να είχαν κράτη όπως η Ισπανία παραδείγματι τη δυνατότητα ε, με την ομοθεσία τους να εξορροπήσουν τις συνθήκες της κρίσης, αλλά δεν κατάφεραν να την αποφύγουν. Τα ρυθμιστικά πλαίσια συχνά θεωρούνται δεσμευτικοί όροι, μέσω οποίου θα πρέπει να δρούν οι επιχειρήσεις. Αλλά με την εξέλιξη που έχουμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα, μάλλον θα πρέπει να μιλήσουμε για αρχές και όχι για κανόνες. Ε, παραθυράκια δε τα οποία επιτρέπουν σε ξένες επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η AAG, η Αμερικανική, ε, θα πρέπει να κλείσουν και θα πρέπει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το συλλογικό όργανο των εποπτών για τις διεθνείς επιχειρήσεις, που όμως δεν ε, εξετάζει επαρκώς την εξάρτηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των ρυθμιστικών τους αρχών από τις εξελίξεις της αγοράς. Είναι πολλοί οι λόγοι που έχω καταγράψει μέσα στην εκθεσή μου. Θα σταματήσω για να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων, εάν με παρακολούθησαν, διότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Και θα ήθελα να ακούσω τι πιστεύετε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ, Κέι. Ε, θα ξεκινήσουμε με την Περβάνς Μπερές, μετά Όλε Σμίτ, ο Σάντζεθ Περσέσο, ο κύριος Αλβαρέθ και ο κύριος Έγκελ. Η Περβάνς έχει το λόγο. Εντυπωσιάστηκα τα μάλα από την ποιότητα της αναλύσεως ε, που έκανε η συνάδελφος και είτε διότι με εξαντλητικό τρόπο εκάλυψε το σύνολο αυτών των ε, θεμάτων, μεγάλη τεχνογνωσία και κάποια σημεία αποτελούν στοιχεία της αναλύσεως που θα πρέπει να κάνουμε και να τα στερνιστούμε και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή. Σωστά υπογραμμίσατε ότι πέρα από το την global imbalance, τη γενική ανισορροπία, τα στοιχεία που αναφέρατε ουσιαστικά δεν είναι τα μόνα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και το θέμα της φύσεως του εσωτερική ζήτηση και εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεως είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Αναφέρατε ότι υπήρχαν καλές και κακές ανισορροπίε. Όταν μιλάμε για ανισορροπίε παγκόσμιες, ο, κα, ο καθένας έχει υπόψη ένα μεγάλο πακέτο Κίνα εναντίον ΙΠΑ. Και όταν βλέπουμε αυτό το μεγάλο πακέτο, τι παρατηρούμε. Αν αυτό το μεγάλο πακέτο επέτρεψε την ανάπτυξη της Κίνας και την έξοδο της Κίνας από την Ένδια, κανείς δεν αμφισβητεί ότι χρειαζόμαστε την, τεκ... την προσωμογή τεκτονικών πλακών τη στιγμή που μπήκε σε αυτόν τον κόσμο η Κίνα των χωρών που ωφελούνται από τα αγαθά της αγοράς. Τι έγινε όμως πίσω από αυτά είδαμε ότι αυτό βασιζόταν σε μηχανισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε αντίστροφα αποτελέσματα. Δείτε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και βλέπετε ότι έχουν εντοπιστεί κίνδυνοι. Οι μηχανισμοί που παρουσιάσατε πράγματι φύστανται. Μα είχε πει κάποιο ότι ουσιαστικά μπορούμε να φανταστούμε ότι οι Αμερικανοί προσπάθησαν να χρηματοδοτήσουν το χρέος του έναντι των Κινέζων. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι και οι Κινέζοι έχοντας επίγνωση του δυναμικού τους, διότι αυτοί βλέπουν μακροπρόθεσμα, και έχοντας επίγνωση τι μακροπρόθεσμε δυνατότητε να ξεπεράσουν την Αμερικανική οικονομία, και βλέποντας ότι όταν ριζοσπαστικά ανέβαν σε ισχύ θα είχαν μεγάλη σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ και θέλανε να ξεφύγουν αυτή τη σύγκρουση και θεώρησαν ότι κατά κάποιο τρόπο καλύτερο θα ήταν να ακολουθήσουν στρατηγική αυτή ισοτιμίας που συνέδεται τα δικά του συμφέροντα με τα Αμερικάνικα συμφέροντα, κάτι που έκαναν μαζικά αγοράζοντα ε, μετοχές αμερικανικές. Παράλληλα από αυτή την αύξηση της ισχύω στα πλαίσια του Global Imbalance, σε παγκόσμιο επίπεδο κανένα μηχανισμός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Παρενέβη στη Γαλλία το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ε, το 69 και το 76 στο Ηνωμένο Ποτέ δεν μπόρεσε να πει τίποτα όμω ούτε για την Κίνα ούτε για τη ΣΥΠΑ. Οπότε αρχές παγκόσμιας διακυβέρνησης και τη έγκαιρη προειδοποίηση που είχαμε δημιουργήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στην πρόκληση ε, δημιουργίας αυτών των τεραστίων ανισορροπιών. Σχόλια. Το μαθηματικό μοντέλο. Αυτά που λέτε είναι κρισίμου σημασίας. Ο πρόεδρος ήθελα συμμετάσχω σε συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων. Τυχαία είναι Γάλλοι αυτοί που αναλύουν το θέμα αυτό ε, των λογιστικών Τι με εξέπληξε από όλα αυτά όμως περισσότερο, από αυτά που συζητήσαμε. Ότι ο πρόεδρος της ACC που δημιουργήθηκε το 1933 άλλαξε το μοντέλο αναφοράς όσον αφορά, που είχε βασιστεί στα αμερικανικά πρότυπα τα λογιστικά για να περάσει ιστορικές τιμές. Μη με ρωτάτε τις θεωρητικές λεπτομέρειες το ζουμί σα λέω από την ανταλλαγή απόψεων που θεωρείς εξαιρετικά σημαντική. Το τέλος του 19ου αιώνα οι μαθηματικοί ξεκίνησαν βασιζόμενοι στο εξή ότι η κατανομή της αβεβαιότητας είναι η ίδια με την κατανομή των σφαλμάτων. Άρα δεν υπάρχει λόγος να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα το θέμα της ιδιαιτερότητας. Και από αυτής της βάσεως έγινε τυποποίηση των λογιστικών βάσει της ε, θεωρίας της σωστής αξίας, σωστής τιμής. Μετά τη μεγάλη κρίση, τη δεκαετία του 20, τέλος δεκαετίας του 20, οι μαθηματικοί αναγνωρίζουν ότι αυτή η θεωρία δεν είναι ακριβής. Και οι οικονομολόγοι ε, ποτέ δεν το δέχτηκαν. Αυτό συνέχισαν να εργάζονται επί μοντέλου που και οι ίδιοι μαθηματικοί θεώρησαν ότι δεν είναι παληθεύσιμο αυτό το θέμα της λήψος υπόψη της αβεβαιότητας στους υπολογισμούς τους λογιστικούς ήταν στο επίκεντρο των ερωτηματικών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της λογιστικής που χρησιμοποίησαμε στο χρηματοστικό σύστημα. Αναφέρεται το θέμα αυτό στην έκθεση. Προτείνω στην έκθεση να πούμε πώς πρέπει να επαναξεταστεί το θέμα αυτό. Δεν θα βρουν τη λύση βουλευτές αλλά πόσο υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά το θέμα της προσαρμογής που απαιτείται. Στα συμπεράσματά σας λέτε κάτι άλλο. Πρέπει να αποθαρρυνθούν οι φορολογήσεις και οι οικονομικές προσεγγίσεις που οδηγούν περισσότερο στη χρέωση παρά στην χρήση ε, αξιογράφων και αυτό μπορούμε να το λάβουμε υπόψη. Όσον αφορά την εσωτερική κατανάλωση στην Κίνα, ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα, αν πάμε και όταν πάμε, να μιλήσουμε και να αναλύσουμε σβάθο το θέμα πάνω σε αυτό. Διότι όπως και η μεταρρύθμιση της υγείας, του τομέα της υγείας στην, στην Αμερική, εξίσου και το δημιουργία συστήματος συνταξιοδότησης στην Κίνα, συμβάλλει πολύ σημαντικά στη δημιουργία αυτής της παγκόσμιας ανισορροπίας της Global Imbalance. Και τέλος, Δεν θα σε εκπλήσω ότι δεν συμφωνώ με τα συμπεράσματά σας όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Πέρα από ε, ήταν οι διάφοροι φορείς ε, βαθμολο... βαθμονόμησης, ε, αξιοπιστίας κάποιων κρατών κλπ. που δαχτυλωτικούνται για την κρίση. Έχουμε παραδείσους που είναι φορολογικοί, εποπτείας και λεύκανσης και αυτοί οι παράδεισοι δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά το διεθνές νομισματικό και χρηματοδοτικό σύστημα. Διότι αυτοί οι τόποι δίνουν προστασία σε χρήμα που ξεφεύγει από την ανακατανομή στις χώρες όπου έπρεπε να γίνει και δίνει την άδεια της δημιουργίας προϊόντων που εκφεύγουν της εποπτείας και των κανόνων, των λογικών και της σωστής διοντολογίας που ισχύουν και ισχύουν στις χώρες που τελικά τα προϊόντα αυτά πολλούνται στους επενδυτές και στους αποταμιευτές. Εκεί διαφωνώ κατά πολύ. Κατά τα λοιπά, πολλές από τις προτάσεις θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτες, τις ενστερνίζομαι και θα, βρουν τη σωστή τους θέση να έκθεση σας υποβάλλω. Ο Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς. Πάντοτε όταν βλέπει κανείς τις σκέψεις του να αντικαταπτρίζονται σε ένα κείμενο με μια καλύτερη διατύπωση, αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά δική μου ερμηνεία και νομίζω ίσως ότι είναι το βασικό συμπέρασμα της Κέι Σφίνμπορν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίω. Και χρειαζόμαστε, και αυτή είναι η δική μου ερμηνεία επιση χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι μετά τι εκλογέ την επόμενη εβδομάδα ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο και η Σουίνμπον, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρα, θα μπορούσε να προσχωρήσει σε αυτέ τι δυνάμει. Εγώ νομίζω ότι σε κάποιο σημείο του εγγράφου που θα γράψει θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία 20 30 χρόνια, το οποίο θεωρώ ήταν ακραία, Γιατί ο κόσμος, ο οποίος τον εγώ ήμουν νεαρός ε, φοιτητής ε, και τον αφέραμε ε, και όταν διαβάζαμε παλιά τον Μάο Τσετούν, αυτά δεν υπάρχουν πλέον και οι άνθρωποι δεν λιμοκτονούν πλέον όπως λιμοκτονούσαν παλιά. Βεβαίως ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στην Αφρική, που ακόμα λιμοκτονούν. Αλλά παρόλα αυτά υπήρξαν τόσα πολλά ευεργετήματα, ωφέλη από αυτή την πολιτική και νομίζω ότι θα πρέπει να το πούμε ρητά. Και αυτό είναι ένα όφελος της παγκοσμιοποίησης χάρη στην παγκοσμιοποίηση συνέβη αυτό και θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά όταν ε, λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να είμαστε σήμερα πιο εθνικιστές και υπάρχουν ορισμένα πολιτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματικά υποφελούνται από τέτοιου ρητορίες. Τώρα, ορισμένες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Και θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό που εξαρτάται από τη, η Κίνα από τις ΗΠΑ και αντίστροφα. Ήταν παράδοξο ότι οι Κινέζοι επέτρεψαν στους ΗΠΑ να καταλάβουν το Ιράκ, να εισβάλλουν στο Ιράκ και να πληρώσουν για τον πόλεμο. Αλλά νομίζω ότι για τους καταναλωτές ήταν εξαιρετικά χρήσιμο όσον αφορά τις χαμηλές τιμές. Και νομίζω ότι υπήρξαν ευεργετήματα και για τους δύο. Και νομίζω επίση ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αναφέρεται εδώ ότι η νομισματική πολιτική δεν ονομάζεται. Εγώ πήγα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, δεν αναφέρεται τον Τόισενμπεργκ, αλλά όταν ο κύριο Τρισέρ ερχόταν για ακροάσει, γινόταν αντικείμενο κριτική για την πολιτική του. Γιατί δεν ε, βλέπετε τι κάνει ο κύριος Γκρίνσμαν. Αυτός είναι που είναι σοφός. Εγώ ήμουν στο γερμανικό στρατόπεδο και δεν το έλεγα, αλλά είναι καλό να το επενθυμίζουμε. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν συνέβαινε πολλά χρόνια πριν. Ακόμα και εδώ στην αίθουσα. Τέλο πάντων, α, δεν θα έπρεπε να λέμε τέτοια πράγματα. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Και επίσης είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση όταν λέτε ότι λόγω ακριβώς αυτής της νομισματικής πολιτικής ε, έπρεπε να υπάρξουν νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιούμε αυτό όταν ασκούμε μια κριτική στον Τρισέ. Και ο Τρισέ πάντοτε έλεγε και ο Ντόζενμερκ επίση, θα μπορούσατε να εξηγήσετε αυτά τα καινούργια εργαλεία. Όχι, όχι στην πραγματικότητα, ούτε καν ε, τα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας. Βλέπετε ότι όλα είναι αλληλένδετα. Και ίσως θα μπορούσατε, ίσως το κάνετε ήδη, αλλά κατά την άποψή μου ε, ενός απλού ανθρώπου, τα τοξικά δάνεια, τα στεγαστικά, στον τομέα των στεγαστικών δανείων, νομίζω ότι έχουμε μια απλή εξήγηση και όταν ε, ε, συναντάμε τους γερουσιαστές θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν εκείνοι οι οποίοι υποχρέωσαν την αγορά των ανυπόθηκων στεγαστικών να είναι τόσο επιθετικοί. Ε, νομίζω ότι από δύο Πομπέι τράγοι μπορούν να βρεθούν ποντού. Αλλά νομίζω πρέπει να το θυμηθούμε ότι ο Μακέιν ήταν νομίζω κάποιος ο οποίος άσκησε τέτοια κριτική, όχι ο παρόν, ο τωρινός πρόεδρος. Και επίση αναφέρεται, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, το έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όσον αφορά τον πληθωρισμό. Ο Στροσκάν είπε ότι αυτό ήταν ένα... Ο Στρασκαν, συγγνώμη, είπε ότι... αυτό ήταν ένα προσωπικό έγγραφο. Ε, νομίζετε πραγματικά ότι είναι μια καλή ιδέα. Ε, κατά δική μου άποψη, γιατί εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου, υποτί... όπου έγινε υποτίμηση του νομίσματος πάρα πολλές ε, φορές. Νομίζω ότι μπορούμε καν να μετρήσουμε πόσες ήταν. Νομίζω ότι η σταθερότητα είναι από τους ακρογωνίους λήθους. Νομίζω ότι αν εγκαταλείψουμε αυτή την ιδέα, αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν αυτό ακριβώς εννοείται ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη σταθερότητα, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο νομίζω επισήμανα ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποια άλλη στόχοι. Αυτά τα... Ε, όσον αφορά τα κριτήρια του Μάστριχτ και τα δάνεια αυτά, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα, μια, ένα ατομικό ποσοστό χρέους, χρέωσης, ε, δημοσίου χρέους για κάθε χώρα. Νομίζετε ότι αυτό θα ήταν σοφό. Δεν ξέρω, έχω πολλούς ενδιασμούς γιατί και αυτό είναι ένα ακρογωνιαίο λίθο σε όλη την ευρωπαϊκή διαδικασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να μα το εξηγήσετε περισσότερο ει βάθο, τουλάχιστον να το καταλάβω εγώ. Αλλά επιτρέψατε μου να καταλήξω λέγοντας το εξή. Δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει ε, κατά ανάγκη να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά τουλάχιστον εγώ το κάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό έγγραφο, πλούσιο σε ρεθίσματα. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω τρία πράγματα για τη διακυβέρνηση, για την νομισματική πολιτική και τέλος για τις ε, παγκόσμιες ανισορροπίες, για τη διακυβέρνηση σε σχέση με το όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, νομίζω και τον τρόπο που θέτουμε τα προβλήματα. Τις τελευταίες μέρες είδαμε πώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το ΕΚΟΦΗΝ και η Κεντρική Τράπεζα εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική κυβέρνηση και στα μέτρα που έχει λάβει για την βελτίωση της κατάστασης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωζώνη επίσης το είπαν. Αλλά ωστόσο η επιστολεπτική, η αξιολόγησης ε, προέβησαν σε περαιτέρω υποβάθμιση. Και νομίζω ότι όλα αυτά θέτουν ε, ζητήματα ε, δεν δίδονται πιστώσεις και από την και ανακύπτουν αυτά τα προβλήματα της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ε, νομίζω ότι το ερώτημα έχει ως εξής. Μπορούν ε, κάποιες ε, κερδοσκοπικές, κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οντότητες, να τηρήσουν τις αρχές της διακυβέρνησης το rating δεν συνιστά απλώ μία γνώμη, είναι μία τοποθέτηση ιδιαίτερω καθοριστική που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τα δικά μας συμφέροντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το θέσουμε αυτό. Το δεύτερο αφορά τη σχέση ιδιωτικού τομέα και δημόσιου τομέα, όπως όλα τα πράγματα. Ε, ε, ο ανταγωνισμός ε, θέτει πολλά προβλήματα εάν νομίζω ότι είναι αναγκαίο να δούμε όλα τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το ζήτημα του ανταγωνισμού και το ζήτημα της ρύθμισης. Τώρα, η νομισματική πολιτική. Εδώ, στο Bretton Woods ε, έγινε μια νομισματική και εμπορική ε, συμφωνία και θεσπίστηκε ένα ενίο. Ε, σύστημα, ούτως ώστε οι πλονασματικές χώρες να μπορούν να χρηματοδοτούν τις ελληματικές ε, χώρες. Αλλά στο Brighton Woods ε, θεσπίστηκε ως ε, σημείο αναφορά στο δολάριο. Η Κίνα κάνει αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη με το δολάριο. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πιο πολυμερή ε, συμφωνία και αυτό προποθέτει μια οικονομική συνεργασία. Γιατί έχουμε και μια αγορά και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες σκέψεις εν σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια βήματα για να βαθύνουμε στην νομισματική πολιτική. Όσον αφορά τις παγκόσμιες ανισορροπίες, θα ήθελα να πω ότι η εξέλιξη ότι σε σχέση με την πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας δημιουργούνται τεράστιες ε, ανισορροπίες. Μέσω της κερδοσκοπίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται. Ε, νομίζω το θέμα της οικονομίας είναι ότι θα πρέπει να χαράξουμε ένα δρόμο ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας και όχι της ονομαστικής οικονομίας. Στην Ευρώπη έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητας το οποίο θέλει να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτή την κρίση είναι ότι εδώ πρόκειται για μια λογική συγκοινωνούν των δοχείων. Και οι δύο τομείς, ιδιωτικός και δημόσιος, τελικά είναι αλληλένδετοι. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά σε μια ευρύτερη προοπτική και να διατυπώσουμε ένα ευρύτερο μοντέλο διακυβέρνησης. Ευχαριστώ κύριε Άλβαρες. Κύριε Άλβαρες. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για την έκθεσή τη και να αναγνωρίσω την πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει, συμπεριλαμβανομένου και του πολύ ενδιαφέροντο σημείου που ξεκινάει τη συζήτηση των επιπτώσεων. Όπως αυτό που συζητήσαμε για την τροποποίηση του ορίου του πληθωρισμού ή την ακαταλότητα του οικονομετρικού προτύπου, την αναγκαιότητα που υπάρχει να βρεθεί ένα καταλληλότερο πρότυπο. Θα ήθελα εγώ όμως να εντοπίσω δύο ζητήματα που έθιξε η συγγήτρια. Τους φόρους για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές καταρχάς, διότι διρωτάται η συγγήτρια εάν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο και αν θα έχει τελικά αποτέλεσμα να περιορίσει τους ε, ε, τις επιπτώσεις χρηματοπιστωτικέ αγορέ. να εξορροπήσει δηλαδή κάπω τι χρηματοπιστωτικέ αγορές. Ναι. Ίσως στην έκθεση να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο φόρος αυτός εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους. Δεν το αναφέρει βέβαια η έκθεση, αλλά σε αυτή τη στιγμή εκδοχή, αλλά ίσως θα πρέπει να το δούμε. Γιατί ένας τέτοιος φόρος και έσοδα εξασφαλίσει και περισσότερη ε, περισσότερο έλεγχο από πλευρά των ευρωπαϊκών οικονομιών στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ε, εξασφαλίζει και σε τελευταία ανάλυση υποχρεώνει το χρηματοπιστωτικό τομέα να προσφέρει και αυτός στην ε, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και επίσης αυτός ο φόρος έχει σαν στόχο να ε, εξισορροπήσει, να αντισταθμίσει τις ε, ε κερδοσκοπικές επιθέσεις και τις συνέπειες τους. Ο φόρος βέβαια πρέπει να είναι διαφανής και η ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα πρέπει να είναι ε, διαφανής. Θα έχει πολύ σημαντική συμβολή πιστεύω ο, φόρο φόρος εάν εισαχθεί. Ένα άλλο σημείο που ανεφέρθη, χωρίς όμως να έχει ε, ιδιαίτερα υπογραμμιστεί, είναι, πιστεύω, ο αγώνας για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι είναι υπέτειοι για την αδιαφάνεια, για την απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων των κρατών μελών. Πρέπει δηλαδή να τους καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους πάση θυσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο Σέγγελ. Το κομμάτι αυτό για τους φορολογικούς παραδείσους που τους λέω εγώ χρηματοδοτικά κέντρα είναι αυτό που μου άρεσε περισσότερο σε αυτά που είπε και η Σουίνμπερν. Ίσως επειδή είμαι Λουξεμβούργιος Όσον αφορά την ουσία να πω κάποια πράγματα. Συμφωνώ με την ανάλυση γενικά. Δηλαδή ότι χρηματοστικά κέντρα μπορεί να είναι, αλλά φορολογική παράδειση δεν είχαν καμία σχέση με τις ρίζες της κρίσης. Μπορούμε να μιλάμε για χρηματοστικά κέντρα για το Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, αλλά όχι για το Λουξεμβούργο, η ρίστα εμπαρόδο. Δεν πήραμε να μιλάμε για την Αγκουίλα, το Ισομάν, το Γιβραλτάρ ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αυτά είναι μέρη όπου περνά το χρήμα. Χρήμα περνά. Και ίσως και αξιόγραφα. Μετοχές δεν δημιουργούνται εκεί. Ποτέ δεν δημιουργήθηκαν εκεί και δεν θα δημιουργηθούν εκεί. Τα προϊόντα που επέφεραν την κατάρρευση του χρηματοπιστικού συστήματος μαγειρεύτηκαν αλλού. Μαγειρεύτηκαν σε ε, μέρη που, που παλιά θεωρήθηκαν, ε, θεωρούνται ότι είναι καλά ρυθμισμένα. Είδαμε πώς ελεγχόταν. Είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά το ρυθμιστικό μας ζήλο. Έχω την εντύπωση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα κατάφεραν να διατηρήσουν κάποια ζωή για την επιδίωξη καλύτερης ρύθμισης, ενώ στην Ευρώπη αυτό που κάνουμε θα μπορούσε και να μην γίνει. Δεν θα κάνει διαφορά. Ούτε καν ασχολούμαστε με τα προβλήματα, ελάχιστα με τα προβλήματα που θα έπρεπε να εξετάσουμε και τα ξαναβλέπουμε ξανά. Δεν είναι καλύτερο έλεγχο, καλύτερη ρύθμιση που θα εμποδίσει αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα τώρα και ίσω συμβούν στην Πορτογαλία αύριο και στην Ισπανία μεθαύριο. Και αν συμβεί και στην Ισπανία, θα συμβεί σε όλη την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη δεν έχει τα μέσα για να σώσει την Ισπανία. Αυτό είναι σαφέστατο. Διότι αν αυτά που συμβαίνουν τώρα πλήξουν μεγαλύτερες χώρες, όλοι θα βουλιάξουμε. Και δεν θα βουλιάξουμε λόγω των οικονομικών κέντρων, των χρηματοστικών κέντρων και των φορολογικών παραδείσων ούτε λόγω κρατικών χρεών δεν θα βουλιάξουμε, αλλά λόγω κερδοσκοπίας, διότι δεν τολμάμε να το αγγίξουμε αυτό το θέμα. Τα θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε και να διερωτηθούμε για αυτά δεν είναι πόσο χρέο είναι λογικό, παρόλο που και αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αλλά το δούμε. Η Ιαπωνία 200% του ΑΕΠ ποσοστό χρέους και δεν έχει χρεοκοπήσει θα μπορούσε να έχει ε, ύφεση για κάποιο, αποπληθωρισμό για κάποια φάση, αλλά δεν έχει χρεοκοπήσει. Δεν είναι τόσο ευάλωτη σε εξωτερικές ε, επιθέσεις και δεν θα χρεοκοπήσει σύντομα. Τελευταία φορά που χρεοκόπησε η Αργεντινή, η Αργεντινή πολλές φορές χρεοκόπησε. 50% το ΑΕΠ είχε χρέος. Όταν η Λετωνία είχε στριμωχθεί, εδώ και κάνα χρόνο, ούτε στο μισό δεν ήταν το επίπεδο του Μάστριχτ για κρατικό χρέος. Δεν υπάρχει αντικειμενικό επίπεδο που θα μπορούσε να προταθεί σε οποιαδήποτε χώρα ή σε χώρες συνδυασμένε, αλλά υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, κακή διακυβέρνηση αιώνια και μας λέγαν ψέματα και κάνανε κολπάκια μας κοροϊδεύαν. Ναι, εντάξει. Αλλά θα μπορούσε η Ελλάδα θεωρητικά να ξεφύγει από εκεί που έχει μπλέξει αν οι αγορές δεν τις έκαναν αυτή, αυτό το έργο αδύνατο. Αν μπορούσε να παγώσει την κατάσταση στην 1η Ιανουαρίου του 2010 και να εφαρμόσει τα σωστά μέτρα θα μπορούσε να είχε ξεμπερδέψει, να ξεφύγει μέσα σε δύο χρόνια. Αλλά τώρα με αυτούς τους ρυθμούς όταν ξαφνικά βλέπεις ότι μόνο για, το, για την εξυπηρέτηση του χρέους πρέπει να επενδύσεις το 50% των δαπανών του προϋπολογισμού και μετά 50% του ΑΕΠ διότι τα επιτόκια ξετρελαίνονται λόγω κερδοσκοπίας, βέβαια κάθε πολιτική δυνατότητα να κινηθεί κανείς από την χάνη Και η Ευρώπη ίσως αποτύχει μάλιστα. Διότι αν αυτό που συμβεί τώρα στην Ελλάδα συμβεί στην Πορτογαλία επίσης και στην Ισπανία μετά ή στην Ιρλανδία μετά Ποιο ξέρει αν δεν συνέβη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν συμβεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Η Ευρώπη θα καταλάβει ότι δεν θα μιλάμε πλέον κατά πόσο η κυρία Μέρκελ συμφωνεί να δώσει μερικά δισεκατομμύρια γερμανικά ευρώ για να δοθούν σε οποιαδήποτε χώρα. Αλλά όλη η Ήπειρος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχουμε αρκετά ευρώ να δώσουμε για τις χώρες. Άρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε να αφήσουμε του φορολογικούς παραδείσους και να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Αυτό που θα πρέπει να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί είναι ότι εντελώς παρανοϊκή, τυχαία συμπεριφορά των αγορών καταστρέφει την κοινωνία στην οποία ζούμε. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό και δεν αντισταθούμε σε αυτό και το αντισταθμίσουμε αυτό, δεν νομίζω ότι θα βρούμε διέξοδο από την κρίση αυτή, την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Σβέν έχει το λόγο. Ε... Ναι, ο Σβέν. Ευχαριστώ. Λέω και Ευχαριστώ πολύ για το έγγραφό σου, Κέι. Ενδιαφέρον, ε, μάλλον, ενδιαφέρον ανάγνωσμα και μάλιστα διότι βλέπω μια παρόμοια προσέγγιση που ακολουθείς για να ανοίξεις κάπως τη σκέψη σου και να εξετάσεις διάφορες πηγές. Αυτό που μου αρέσει πολύ, παραδείγματος χάρη, είναι σαφής δήλωση ότι δεν μπορείς να σπάσεις φυσαλίδες φούσκες με νομισματική πολιτική, διότι πολλοί το διατείνονται αυτό. Το άκουσα συχνά εδώ στην Επιτροπή. Για να αποφύγουμε τις ε, φούσκες αυτές, τις φυσαλίδες όπως τις είδαμε, πρέπει να αυξήσεις αρκετά τα επιτόκια αλλά μετά δεν σου μένει πολύ από την πραγματική οικονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ ισχυρό σημείο. Λόγω περιορισμένου χρόνου έχω να αναφέρω μόνο δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα η πηγή της κρίσης, το αίτιο της κρίσης και κάποια μακροοικονομικά στοιχεία. Οι βασικοί λόγοι για τη ρευστότητα... Α, εδώ λείπει μια πτυχή όσον αφορά το θέμα. Λόγω παγκοσμιοποίησης, το μερίδιο του εργατικού δυναμικού στο ΑΕΠ, η αμοιβή του εργατικού δυναμικού ε, μειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό προσέθεσε στην ανισότητα. Και αυτή η πρόσθετη ανισότητα διότι αν έχεις μεγαλύτερο μερίδιο που πάει στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, τότε θα έχω μεγαλύτερη τάση να αποταμιεύουν. Και αυτό τροφοδοτεί επιπλέον τις άλλες πηγές ρευστότητας που ανέφερες. Έχω την εξής εντύπωση. Κανονικά η πολιτική αριστερά λησμονεί τις, νομ... νομισματικές πολιτικής πολιτικές, τις πηγές πολιτική για την ρευστότητα και η δεξιά ξεχνά την ανισότητα και αυτό δεν μ' αρέσει. Αν σκεφτούμε αυτές τις, αυτή την πηγή της ανισότητας και το δούμε σαν παγκόσμιο φαινόμενο, τότε μπαίνει στην εικόνα και η φορολόγηση. Γιατί, διότι αν έχεις πρόβλημα λόγω μείωση των διαπραγματευτικών δυνάμεων του εργατικού δυναμικού λόγω παγκοσμιοποίηση, θα μπορούσε να έχει φορολογικό σύστημα για να επανεξισορροπήσει την κατανομή. Και τότε έρχεται ο φορολογικός ανταγωνισμός. Επειδή υπάρχει ανταγωνισμός όχι μόνο μεταξύ διαφόρων περιοχών και εργαζομένων εργατών, σε διεθνέ επίπεδο, αλλά και μεταξύ φορολογικών συστημάτων, τα οποία φορολογικά συστήματα υποτίθεται ότι είναι το πλαίσιο τη οικονομία αγορά και αποτελούν τμήμα του πλαισίου τη οικονομία αγορά, με, με την καλή έννοια του γερμανικού όρου Ordnungspolitik, ε, τότε έχει πρόβλημα. Διότι το σύστημα που υποτίθεται ότι επανεξισορροπεί και διορθώνει τις, τα προβλήματα της αγοράς, τα κενά της αγοράς, δεν μπορεί να καθοριστεί δημοκρατικά πλέον, αλλά από μόνο του ε, μπαίνει σε ανταγωνισμό και είναι πολύ περιορισμένο το τι μπορεί να κάνει. Και εδώ ξαναμπαίνει το Λουξεμβούργο στην εικόνα, πρέπει να το πω αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό οικονομικό ζήτημα. Η έλλειψη δυνατότητας επανεξισορρόπησης της αύξησης ανισότητας μέσω φορολόγησης, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Και θα πρέπει να εξεταστεί στην Ευρώπη, να το εξετάσουμε και διεθνώς. Και αυτό που δεν μ' αρέσει και σε κάποιες φάσεις το έγγραφο χάνεται είναι ότι αυτά μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να τα εξετάσουμε, διατείνεται. Δεν το πιστεύω αυτό. Το παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να εξετάζεται και δεν μπορεί να έχεις ατέρμονες ρυθμίσεις μόνο στην Ευρώπη και πουθενά αλλού, αλλά μπορεί να κάνεις αρκετά πολλά στην Ευρώπη, διότι εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλη αγορά, να ρυθμιστεί από πολλές πλευρές. Γι' αυτό, για μακροοικονομικούς λόγους, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, τελευταίο μου σχόλιο αυτό, η κοινωνική κρίση. Αυτή η κρίση, αυτή η επιτροπή, συγγνώμη, δεν ονομάστηκε ε, μόνο επιτροπή για την χρηματοστική κρίση, αλλά και για την κοινωνική κρίση. Αλλά στην ανάλυση σου για το φόρο δεν το ανέφερες. Θα, εδώ θα πρέπει τι λες εδώ, ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη τελικά, πρέπει να φορολογήσουν τους λαούς τους και αν καμιά φορά αποταμιεύεται πλούτος σε φορολογικούς παραδείσους, τότε η φορολόγηση μετακινείται χρονολογικά. Όχι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι συνέπειες των επιτοκίων είναι πολύ σημαντικές. Αν δεν πληρώνεις για 20 χρόνια και φορολογεί 20 χρόνια μετά, κάνει τεράστια διαφορά όσον αφορά το ποσό που φορολογεί για κοινωνικούς λόγους. Εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την μη φορολόγηση κεφαλουχικών εισοδημάτων και πλούτου σε κάποια μέρη και τις μη δυνατότητες εφαρμογής του φορολογικού δικαίου, εθνικού φορολογικού νομ, ε, νομολογίας. Κυρίως αν θες να υπερασπιστείς την κυριαρχία τη φορολογική των κρατών μελών. Πρέπει να είναι κανεί κατά τη δυνατότητα πλούτο να μετακινείται και να πηγαίνει αλλού και να αποθηκεύεται. Και υπάρχει ασυνέπεια στη φιλοσοφία αυτή, όπω την αντιλαμβάνομαι εγώ, όσο αντιλαμβάνομαι τη θέση του κόμματό σου για την ε, οικονομική πολιτική. Απ' τη μία λες ότι είναι εθνικό δικαίωμα φόρος και από την άλλη υπερασπίζεσαι την ίδια δομή που υπονομεύει αυτή την ε, ε, κυριαρχία. Και εκεί έχει σοβαρέ ελλείψει στο έγγραφό σου που ριζώνει σε κάποια πεθυθήσεις κατά την άποψή μου παρά σε σαφή ανάλυση αυτή η προσεγγίση σου. Έχουμε πολύ... Έναν πολύ γνωστό προσκεκλημένο. Ο κύριος Μέισιν ήρθε στην Επιτροπή μας. Πρώην μέλος της Deutsche Bundesbank, της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, έχει συζήτηση τώρα το μεσημέρι με τους συντονιστές της Επιτροπής μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε ευχαριστούμε που μας ε, δίνετε λίγο περισσότερο χρόνο από το χρόνο σας και έρχεστε και στην ολομέλεια της Επιτροπής μας. Να ακούσουμε τον κύριο Χούντι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι άκουσα με προσοχή την παρουσίαση της έκθεσης που έκανε η συγγήτρια. Διάβασα το κείμενο που μας έχει μοιραστεί και την ευχαριστώ πολύ. Όπως επίσης ευχαριστώ πολύ και για το αναλυτικό κείμενο που είχε την καλοσύνη να μας μοιράσει και υπόσχομαι να το μελετήσω με, με σοβαρότητα και με, ε, με προσοχή. Συμφωνώ με την κριτική που ασκεί το κείμενο και η συγκήτρια στα μαθηματικά μοντέλα που ακολούθησαν οι τράπεζες όσο αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής. Όμως, πρέπει να πω ότι σε βασικά σημεία της ανάλυσης στα θέματα που αντιμετωπίζει και στις κατευθύνσεις και στις προτάσεις που κάνει δεν συμφωνώ. Ε, και με αυτή την έννοια θα πω κωδικοποιημένα ποιε είναι η διαφορετική αντίληψη στα ζητήματα έτσι όπως τα αντιμετωπίζει το κείμενο και η συγγήτρια. Στο πρώτο, μιλάει για <clears throat> ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία. Η αντίληψη του κειμένου ότι αυτές οι ανισορροπίες οφείλονται σε λανθασμένε λανθασμένες πολιτικές ή αρνητικές διακρατικές, αρνητικούς διακρατικούς ανταγωνισμούς, δεν νομίζω πως αποδίδει την πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, οι ανισορροπίες στο παγκόσμια οικονομία, στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, αυτό δεν είναι το σύστημα, είναι δομικού χαρακτήρα. Στο τέλος τέλος, τι είναι, έχουμε έναν ανταγωνισμό κεφαλαίων Εντό εκτό των συνόρων μιας χώρας και έχουμε και ανταγωνισμό κεφαλαίου και εργασία. Αυτό είναι παραδεκτό, αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό. Αυτοί οι ανταγωνισμοί δημιουργούν ανισορροπίες, δημιουργούν κρίσεις. Ε, ένα παράδειγμα, τα πλεονάσματα στις χώρες που αναφέρονται, στην Κίνα, στη Γερμανία, δεν οφείλονται σε ακραίο μισθολογικό ντάμπινγκ που έχουν ακολουθήσει αυτές οι χώρες τηρουμένων των αναλογιών. Αυτό το στοιχείο παρακάμπτεται. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πλέον έθματα. Δεν υπάρχουν και αυτές οι αιτίε. Δεύτερο, στη νομισματική πολιτική. Συζητούμε για τα χαμηλά ή όχι επιτόκια. Είναι γεγονός ότι τα χαμηλά επιτόκια οδήγησαν στις Ηνωμένε Πολιτείες και αλλού στη φούσκα των ακινήτων. Όμως, ποιος τίναξε το παιχνίδι στον αέρα. Δεν ήταν η οχι επιτοκια ειναι γεγονος οτι τα χαμηλα επιτοκια οδηγησαν στις ΗΠΑ και αλλου στη φουσκα των τραπεζών, των κερδοσκόπων, που μπήκαν σε αυτές τις υποθέσεις και το τίναξαν, τίναξαν όλη αυτή την υπόθεση στον αέρα, διότι είχαμε μια υπερεκτίμηση, υπερδραστηριότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα που παρέκαψε για κάποια στιγμή ίσως το ίδιο αυτό καθ' αυτό το χρηματιστήριο και μπήκε μέσα στην αγορά των ακινήτων και στα στεγαστικά δάνεια και στην ασφάλιση αυτών των ακινήτων. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι μόνο το παιχνίδι με τα επιτόκια, είναι και πώς λειτουργεί και με κάτω από ποιου όρου και κάτω από ποιο έλεγχο. Τολμώ να πω το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο τρίτο, μαζί με άλλου συναδέλφου, δεν συμφωνώ με την ανάλυση που κάνει και τον τρόπο αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων. Πρέπει να υπάρξει ένα να αντιμετωπιστούν. Δεν νομίζω ότι προσφέρουν. Σε κάθε περίπτωση έχουμε κάνει και αναλυτική συζήτηση. Ε, ένας φόρος επί των συναλλαγών ενδεχομένως θα περιόριζε την ασυδοσία ε, μάλλον θα περιόρισε το μέγεθο του χρηματοπιστωτικού τομέα, που επαναλαμβάνω ότι ένα από τα σημεία τη κρίση, κατά την άποψή μου βεβαίω, είναι η υπερδιόγκωση, η υπερδιόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα σε δραστηριότητε που δεν το ανήκουν, θα έλεγα κατά μία έννοια, ή που έτσι όπω μπήκε και με αυτόν τον τρόπο και με την ασυδοσία, κατάφερε να οξύνει αρκετά προβλήματα της, ε, της κρίσης. Και η τελευταία μου παρατήρηση, μιλάμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση και τα προβλήματα και τι πρέπει να γίνει και δεν ξέρω βεβαίως αν είναι αντικείμενο του ιδίου του κειμένου, αν είναι αντικείμενο σίγουρα της συνολικής μας έκθεσης, να κάνουμε μια αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν από τους θεσμούς ως μορφής διακυβέρνησης. Ήδη ε, οι συζητήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο και έχουν αφορμή την Ελλάδα, διαβάζω τώρα σήμερα χτες, αρχίζουν περισσότεροι πλην ορισμένων να διαπιστώνουν το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Τι φταίει. Γιατί η Επιτροπή, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χειρίστηκαν έτσι τα θέματα και κατέληξαν. Καταλήγουμε σήμερα να έχει οδηγηθεί η Ελλάδα, χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, στις δαγκάνες θα πω εγώ, στα πλοκάμια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό δεν είναι πρόβλημα ρύθμιση, δεν είναι πρόβλημα διακυβέρνηση, δεν είναι πρόβλημα σχεδιασμού, δεν είναι πρόβλημα προοπτική. Νομίζω υπάρχουν, επιτρέψτε μου δύο κουβέντε, υπάρχουν οι ελληνικέ ιδιομορφίε, οι ελληνικέ ιδιαιτερότητε. Προσυπογράφω το κατηγορό που έχει αποδοθεί σε σχέση με την εικόνα τη ε, ελληνική οικονομία, τη ευθύνη των κυβερνήσεων. Άλλωστε δεν έχω και κανένα λόγο. Αλλά όπω βλέπετε, μέρα τη μέρα διαπιστώνουν το πρόβλημα είναι γενικότερο. Θέει διαφθορά στην Ελλάδα, τα λάθο στοιχεία που εδίδονται. Μα ήταν, έχουμε και χώρε που έδιναν σωστά στοιχεία, αλλά δεν απέφυγαν τα σημερινά προβλήματα και επομένω πρέπει να τοποθετηθούμε, να τοποθετηθούμε, να κάνουμε μια εκτίμηση. Ξαναλέω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω μορφή διακυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, πώ έχει θεμελιώσει την, οικονομική, την νομισματική πολιτική, τι σημαίνει ο μηχανισμό του ευρώ, τι σημαίνουν τα δομικά κατά την άποψή μου κενά, γιατί αυτό ο μηχανισμό δεν προέβλεπε, δεν έχει μηχανισμό αντιμετώπιση κρίσεων και είδατε που φτάσαμε στα, στις δαγκάνες του Διεθνούς και άλλες πλευρές που αξίζει τον κόπο νομίζω να κουβεντιάσουμε. Επομένως θα έλεγα ε, ναι, συζητάμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση, ας δούμε όμως και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μορφή διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χουντή. Υπάρχουν δύο ακόμα παρεμβάσεις και στο τέλος θα δώσω συντομία το λόγο στην κυρία Σφίνμπορν. Η Ντονάτα Χίμπνερ έχει το λόγο. Thank you uh, very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ έκανα κάποιες σκέψεις ε, γιατί βρίσκω τόσο καλή την έκθεση της ΚΕΙ και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι την εκτιμώ γιατί πραγματικά αναφέρεται, θίγει ε, σημαντικά στοιχεία της νέας παγκόσμιας ε, κρίσης. Διαβάζω αυτή την έκθεση σαν μια προσπάθεια ε, εντοπισμού αυτών των στοιχείων, ε, μιας νέας κατάστασης που εμφανίζεται ως φυσιολογική. και θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα στοιχεία που αφορούν αυτούς τους νέους, μάλλον τους νέους κανόνες ότι πρώτον είναι το κεφάλαιο θα είναι πιο δαπανηρό στο μέλλον. Οι Αμερικοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα μετατρέπουν σε μια οικονομία αποταμιευτών και ίσως και η Κίνα ε, θα μετατραπεί σε μια οικονομία καταναλωτών. Αυτή είναι μια νέα νόρμα. Τώρα, το θέμα μου είναι πού θα βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός αυτής της ε, Θα υπάρξει μια νέα ισορροπία ή ανισορροπία. Ε, θα, θα, που θα διηγηθούμε μέσω της ιδιαίτερης μας πολιτικής ε, και στρατηγικής. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Αμερική που επιφελήθηκε τόσο πολύ από τις χαμηλές ε, τιμές της Κίνας, αλλά και η Ευρώπη, όπου, νομίζω, όπου θεωρώ ότι είχαμε ε, πολύ, είχαν πολλά πλεονεκτήματα από τις, πολλά από τις χαμηλές τιμές της Κίνας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το μέλλον εν σχέση με το πού τοποθετείται ακριβώ η Ευρώπη και τι είδου πολιτική θα πρέπει να χαράξει η Ευρώπη για να βρει τη σωστή της θέση εντός αυτής της νέας παγκόσμιας συγκυρίας και κατάστασης. Νομίζω αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η ανάδυση αυτή της, ε, των νέων μετακρίση ε, κανόνων ε, σημαίνει ότι δεν θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις σε μια ανοιχτή οι προκλήσεις θα γίνουν τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να υπάρξει μια σταθερή πρόοδος ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την περαιτέρω βελτίωση των ρυθμίσεων. Αλλά για να αποφύγουμε και οι τοπαθείς τάσεις, ε, όπως ε, τάσεις προστατευτισμού κλπ και φοροδιαφυγής σε φορολογικούς παραδείσους. Νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ίδια μας τα συμφέροντα ε, στο μέτρο που τα ελλείμματα πραγματικά περιορίζουν τις δυνατότητές μας οικονομικής μεγέθυνσης, ανάπτυξης. Νομίζω ότι το καθήκον μας θα είναι ε, να προαγάγουμε ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο θα ανταμείβει ένα ανοιχτό σύστημα για στρατηγικές που προέρχονται από την αγορά και αυτή η ανοιχτή μορφή της παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει νομίζω να κατοχυρωθεί στην διαμόρφωση, στην εκπόνηση αυτού του νέου συστήματος. Ε, το σύστημα εμπορίου θα πρέπει να επιβιώσει μέσω βεβαίω όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά την ανάγκη να έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο να λειτουργεί με έναν βιώσιμο τρόπο, αηφόρο τρόπο, όχι μόνο για ένα χρονικό διάστημα, αλλά για τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί εάν το μεταρρυθμίσουμε κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τις ανησυχίες ή τους φόβους των περισσότερων συμμετεχόντων του παγκόσμιου παιχνιδιού όλους τους ενεχόμενους, αλλά και τις φτωχές ε, αναπτυσσόμενες χώρες γιατί νομίζω ότι η εμπειρία μας δείχνει ότι εάν τα ενδιαφέροντα κάποιου δεν λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο ενός σφαιρικού μοντέλου συστήματος, ε, νομίζω ότι αυτό θέτει τεράστιες προκλήσεις σε όλους όσους μένουν απ' έξω ή έχουν αυτή την αίσθηση. Το τελευταίο σημείο είναι το εξή. Εάν διάβασα στην την έκθεσή σα, λέτε και συμφωνώ μαζί σα, το πώ το νέο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ε, ε αυτό μένει ε, να το δούμε, γιατί βρίσκεται υπό εξέλιξη. Αλλά όσον αφορά αυτό το νέο σύστημα ε, και τα αδρά του χαρακτηριστικά, νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ειδικά σήμερα όπου γνωρίζουμε τους κινδύνους της ε, χρηματοπιστωτικής οικονομίας και της εθνικής υπερχρέωσης. Εάν θέλουμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, νομίζω ότι τα αδρά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος θα συνοψίζονται στην δυνατότητα να συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη και να παράσχει τα κατάλληλα εργαλεία για αποταμιεύσεις και παρά το ακριβό κεφάλαιο ε, χρηματοδότηση, να παράσχει χρηματοδότηση στην ανάπτυξη. Και για να καταλήξω, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να στοχεύσουμε σε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ ε, ρίσκων και τίμηση ρίσκων και ανάπτυξης. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προέλθει από τις παρούσες ε, μεταρρυθμίσεις. Κύριο σας ευχαριστώ πρόεδρε που μας σύντομο κι εγώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω, εάν μου επιτρέπετε, δύο-τρία πράγματα. Καταρχάς για την έκθεση. Από την έκθεση αυτή, νομίζω ένα από τα σοβαρότερα συμπεράσματα είναι το σχετικό με το ρόλο των ε, ε, φορολογικών παραδείσων στην κρίση. Και ακούμε να, γίνονται, να γίνεται συχνά λόγος για την κερδοσκοπία όλο και περισσότερο και κάποιοι προσπαθούν ε, να εκμεταλλευτούν ε, την αύξηση των επιτοκίων των κρατικών, του κρατικού χρέους διαφορών κρατών. 75% των hedge funds έχουν, είναι σε χαρτοφυλάκια μέσα στους φορολογικούς παραδείσους. Δεν μπορείτε να μας λέτε λοιπόν ότι δεν έχουν ρόλο στην κρίση φορολογική παράδοση γιατί ψωτα δεν αληθεύει αυτό. Ρύθμιση και έλεγχος δεν υπάρχει. Και γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη τέτοια ε, την ανάγκη όταν δίνονται τέτοιου είδου πληροφορίε, εμεί ω φιλελεύθεροι τουλάχιστον, γιατί δεν είμαστε κατά του έλεγχου, έλεγχου τη αγορά, ναι, ίσω ο κύριο Σμίτ, αλλά 75% δεν μπορεί να μείνει έξω από τον έλεγχό μα, έξω από τον έλεγχο των κρατών. Και επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό, η δυνατότητα για χώρες μεμονωμένες στην ε, ε, ασφαλισμένες σημεία, αλλά πάντως βρίσκονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ελέγχονται από τα ευρωπαϊκά όργανα, από, τις, ε, από τα ευρωπαϊκά κράτη, από κάποιον ευρωπαϊκό θεσμό. Ε, ετέθηκε το ζήτημα και μέσα στην έκθεση της ΑΕΚΕ. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε και υπό αριθμόν 3 πρέπει να βάλουμε και κάτι το θετικό με στην έκθεση. Το θετικό είναι ότι δεν αντιμετωπίσαμε περίπτωση αντίστοιχη με αυτή των Lehman Brothers. Και θυμάμαι στα τέλη του 2008 πώς είχε ακουστεί μία σχετική νήξη. Πολλά ήταν τα προβλήματα. Πολλά από τα χρήματα του φορολογούμενου είχαν, και με συγχωρείτε που το λέω, ξεκινήσει από τη Γερμανία ή από τη Λετωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο να επενδύονται στις κάτω χώρες αλλά φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαμε διασώσει τις τράπεζες και είχαν χαθεί όλα αυτά. Όλα Υπήρχαν πολύ πιο σοβαροί φόβοι από αυτά που τελικά είδαμε να συμβαίνουν. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει και με την ε, οικονομική διακυβέρνηση μέσα στην Ευρώπη. Δεύτερον και τρίτον, έχοντας περάσει κάποιες εβδομάδες στις ΗΠΑ πρόσφατα και έχοντας προσπαθήσει να μάθω από πρώτο χέρι ε, τις πληροφορίες, ο κύριος Πόσον, όπως ξέρετε, είχε πρώην ε, υπουργό των οικονομικών, ε, του, του, Treasury δηλαδή των ΗΠΑ, ε, είχε γράψει ένα βιβλίο για την κρίση, με τις προβλέψεις για την κρίση. 55 εκατομμύρια ήταν οι υποθήκες που κατέρευσαν στις ΗΠΑ. πολιτειες Πολιτείες. 13-3 εκατομμύρια και ο κύριος αυτός έλεγε ότι τα 7 εκατομμύρια ήταν λίγο πολύ απολεσθέντα δάνεια. 1,4, 1,6 ίσως 3 εκατομμύρια δολάρια. Και κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει με το εμπορικό δάνειο για την, με τις εμπορικές υποθήκες. Αυτά που μιλάμε είναι μόνο τα στεγαστικά. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι η κρίση αυτή έχει εισαχθεί στην Ευρώπη. Είναι η εισαγόμενη κρίση. Και αν κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά, ναι, δεν έχουμε προστατέψει εαυτούς. Εάν δούμε τις, Ευρω... τις Αμερικανικές τράπεζες πώς χειρίστηκαν την υπόθεση, αν δούμε τα ισοζυγιά τους και ένα εσωτερικό εγχειρίδιο πρέπει να σας πω ότι αναφερόταν στις ΗΠΑ για τη Lehman Brothers και φάνηκε ότι όταν άρχισαν ξαφνικά την, ε, την πίεση αυτή οι τιμές υπήρξε μία προσπάθεια επιτυχής εν τέλει να πιεστεί, να συμπιεστεί η κρίση και να εξαχθεί στην Ευρώπη. Και αυτό το κάνανε χάρη στους ολογισμούς των επιχειρήσεών τους. Και αν δείτε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα αρχίζουν πάλι να χορηγούν δάνεια, αρχίζει μια νέα δραστηριότητα. Στην Ευρώπη αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς είναι το ερώτημα του ποιες πόσες είναι οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις που έχουν συμπιεστεί κατά αυτόν τον τρόπο και έχουν εισαγάγει την κρίση. Θα το δούμε ίσως και αυτό. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές, ότι δεν έχουμε προστατέψει αυτούς από την εισαγόμενη κρίση. Για διάφορους λόγους. Την επόμενη φορά όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ. Οκ. mm. κάναμε τη χάρη. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό περνώντας αρκετό χρόνο σε αυτή την έκθεση ότι βλέπω ότι το διάβασαν συνάδελφοι και είμαι ευγνώμων που χρησιμοποίησατε το χρόνο για να το δείτε και ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια που ακούστηκαν. Να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία που αναφέρθηκαν και θεωρώ ότι σημαντικό ένα έγγραφο όπως αυτό να είναι ένα επίμαχο έγγραφο. Δεν περίμενα να συμφωνήσουν όλοι με τα πάντα διότι και πολλοί από το κόμμα μου δεν θα συμφωνούσαν με όσα περιέχει το έγγραφό μου. Το πιο επίμαχο σημείο αφορούσε το έγγραφο του Ιθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχω μεγάλο σεβασμό για την για τον Λίβιε Μπλανσάρτ και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απορριφθεί η έκθεσή του να θεωρηθεί προσωπικό έγγραφο. Πιστεύω ότι ο στόχος του 2% ε, πληθωρισμό ε, είναι παλιό στόχος για πολλά χρόνια και να πούμε ότι δεν αλλάζει αφού άλλαξε ο κόσμος στις τελευταίες δύο δεκαετίες ε, ίσως να μην είναι σωστό. Ίσως πρέπει να αναλύσουμε ποιο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο. Ίσως 0,5% ένα 0,5% δεν θα έκανε μεγάλη διαφορά ε, στην παγκόσμια οικονομία να μας έδινε κάποια δυνατότητα ελιγμού στην κρίση. Δεν ξέρω, απλώς αισθάνομαι ότι χρειάζεται κάποια ανάλυση, κάποια συζήτηση και ίσως να ήταν κάτι υγιές. Δεν θα ήθελα το εγγραφό του να πεταχτεί στα σκουπίδια με τη μία. Δεν συμφωνώ, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση. Είναι σημαντική όσον αφορά τώρα το ΑΕΠ και το ποσοστό αυτό ΑΕΠ έναντι χρέου και τα κριτήρια του Μάστριχτ. Και εδώ υπάρχει κάποιο επίμαχο σημείο. Παίζω το δικηγόρο του διαβόλου, δεν ανήκω στην Ευρωζώνη και ίσω είναι άδικο που το κάνω αυτό. Αλλά τα ποσοστά δεν τηρήθησαν στη χώρα μου και στα περισσότερα άλλα κράτη-μέλη. Και ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί και ίσως αυτές τις συμφωνίες στα κράτη-μέλη να τα ρυθμίσουν σε αυτό που ήταν καλό για την Ελλάδα να μην ήταν καλό για τη Γερμανία. Ίσως χρειαζόταν περισσότερη ανάλυση, λεπτο, μικρορύθμιση. Δεν λέω ότι κάθε κάτω μέλος θα έπρεπε να ρυθμίζει αυτό, αυτά τα ποσοστά, αλλά να αναλύουμε τις αναλλακτικές λύσεις και αν δεν λειτουργήσε το ένα ποσοστό, ίσως θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ε, και εμπειρογνώμονες να δώσουμε μια αναλλακτική λύση. Πρέπει να πω ότι υποψιάζομαι ότι υπερβάνς και ο Σβέν και άλλοι θα με βρουν σύμφωνοι όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Το συζητήσαμε επανειλημμένα πολλές φορές και πραγματικά θεωρώ, πιστεύω ότι υπάρχει ένας λόγος όπου το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ φοβούνται λιγότερο του φορολογικού παραδείσου. Οι μεγάλε επιχειρήσει χρησιμοποιούν περισσότερου φορολογικού παραδείσου για διάφορο, διάφορα προϊόντα χρηματοστατικά διότι έχουμε και για σε ατομικό επίπεδο και σε εταιρείε ε, φορολόγηση εισόδων. Ε, και αν δεν το αποκαλύπτεις ότι πας σε φορολογικό παράδεισο, διαπάτης αδίκημα και το κάνεις. Ε, υπάρχουν φορείς για φορολογική ε, ουδετερότητα και στην Οικονομική Επιτροπή θα τα συζητήσουμε τα θέματα και θα γίνουν μάχες και περιμένω πώς και πώς. Σας ενθαρρύνω όμως να πάτε στις νήσους Κεϊμάν και να δείτε πόσο ρυθμισμένη είναι αυτή η αγορά των ίσων και ημάν. Δεν είναι αρρυθμιστή και αν κάποιος διατείνεται ότι δεν ξέρουν τι κάνουν και ότι δεν το εξετάζουν, πηγαίνετε να επισκεφτείτε να διαμορφώσετε γνώμη. Υπάρχουν πολλά μέτρα, πολύ ρυθμισμένη αγορά, ε, και είναι άδικο να λέμε ότι το κάνω Όσον αφορά το τι καλύπτει η έκθεση, πραγματικά να ε, παραδέχομαι ότι φτάσει σε σελίδε είναι δύσκολο καθήκον. Προηγήθηκαν πολλέ εκθέσει που συζήτησαν πολλέ από τι κοινωνικέ πτυχέ και θεώρησα ότι να εστιαστώ στο χρηματοδοτικό τομέα και στα οικονομικά αίτια ίσω ήταν το σωστό που θα έπρεπε να κάνω, αλλά να γνωρίζω και παραδέχομαι ότι υπάρχουν κάποιε ελλείψει και νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά κενά και ελλείψει. Αλλά δοθέντω του χρόνου και όλων των άλλων περιορισμών, εστιάστηκα ε, ε, σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πεδίο και η λειτουργήσε υπέρ μου. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που το διαβάσατε το έγγραφο και τα σχόλιά σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Αυτό είναι το τέλος της πρωινής συνεδριάσεως, των πρωινών συνεδριάσεων, το απόγευμα, στις 3 η ώρα το απόγευμα, έχουμε παρουσίαση της Copenhagen Economics, της αξιολογής των συνεπειών όσον αφορά της, των δράσεων που δεν είναι παρκώς συντονισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της κρίσης. Περιμένω να δω τους περισσότερους από εσά εδώ παρόντες το απόγευμα. Καλή σας όρεξη.